Κυρίες και κύριοι, έχουμε απαρτία. Σας καλωσορίζω στην πρώτη μας συνεδρίαση μετά την αλλαγή της χρονιάς. Εύχομαι σε όλους ένα αίσιο και ευτυχές και επιτυχές νέο έτος. Παρακαλώ να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι, πιο υγιείς από μένα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο χιονιά στη Γερμανία και έχω κρυολογήσει. Όταν έχει χιόνι πρέπει να καθαρίσει και όλα αυτά και έχω ξεσυνηθίσει σε όλα αυτά. Ερχόμαστε τώρα στην ημερήσια διάταξη, την έχετε, δεν έχει ζητήσει κανεί καμία αλλαγή, δεν ξέρω να υπάρχει επιτυχία, επιθυμία, συγγνώμη. Ε, Σημείο 2. Έχουμε το Cont News με τις διάφορες γλώσσες που ε, υπάρχει διερμηνία και επίσης ε, η ε, συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Έχουμε ψηφοφορίες τώρα. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες στα μηχανήματα. Έχουμε βέβαια και κάποιους απόντες λόγω καιρού λόγω της κακοκαιρίας. Παρ' όλα αυτά δεν θα περιμένουμε γιατί είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Ε, θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για το πολιτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη συνθήκη. Ε, ο κύριος Στεχόφσκι είναι εισηγητής, ο οποίος δεν θα λάβει το λόγο διότι είναι απόν. Είναι έτοιμες οι πολιτικές ομάδες να ψηφίσουμε, παρακαλώ. Η τροπολογία υπαριθμών 3 ψηφί Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά Παρακαλώ, σηκώστε ξανά τα χέρια σας. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ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 Η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στο σύνολο της τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Πέρας. Ομόφωνα. 8 ψηφί υπέρ με 8 παρόντες. Yeah, Dann bitte die andere Maschine nehmen. Ja, danke. Παρακαλώ, αλλάξτε μηχάνημα αν δεν λειτουργεί το μηχάνημά σα. Ε, το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Κοινή δήλωση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Δεγιόνκ. Επιθυμεί το λόγο. Όχι. Ωραία. Και περνούμε στην ψηφοφορία. Η τροπολογία 1. Ψηφί Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην ονομαστική τελική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα, παρακαλώ. Πέρασε. Οχτώ ψήφοι υπέρ και δύο εποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κυρίου Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ. Και προχωρούμε. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Συνεχίζουμε το σημείο 5 στη μέση διάταξη για την Χρηματοδότηση. Α, ποιος εκπροσωπεί την κυρία Κλάουδια Σμιτ, την εισηγήτρια. Er Έχει δει κανεί τον κύριο Τσέλερ. Ε, υπάρχει κανένα συνεργάτη του εδώ. Η κυρία Σμιτ μα ανακοίνωσε, κοινοποίησε ότι κολλείεται έχει αποκλειστεί στην Αυστρία από την κακοκαιρία και ο συνάδελφος Τσέλερ την εκπροσωπεί. Χτες μας είπαν ότι ε, ε χτες απείλησαν με απεργία στο Βερολίνο και σήμερα απήργησαν. Δεν ξέρω τώρα να περιμένουμε τον εισηγητή. Ο κύριο Σαλαφράγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι το εξή διευκρινιστικά. Έκανα λάθος την προηγούμενη ψηφοφορία. Ήθελα να υπερψηφίσω την τελευταία νομοδότηση την κοινή δήλωση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των αποκεντρωμένων ε, ε, οργανισμών. Έκανα λάθο και παρακαλώ ε, να αλλάξετε, μάλλον να μην ληφθεί υπόψη η θετική μου ψήφος. Μάλιστα, θα το σημειώσουμε. Τώρα τι έγινε με τον συνάδελφο. Έρχεται σε ένα λεπτό. Ο αναπληρωτή της εισηγητρία. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε μπει ακόμα σε ρυθμου δουλειάς. Σιγά σιγά.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 Λοιπόν, είμαστε στο σημείο υπαριθμών 5 τη ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για μια γραμματότηση που αφορά στη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση τη κοινή γεωργική πολιτική. Ε, και έχετε παρακαλώ το λόγο για να μα μεταφέρετε την άποψη τη εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας εύχομαι καλή χρονιά. Σε εμά στο Βερολίνο τα πράγματα ξεκίνησαν ε, με απεργία στο αεροδρόμιο, σε τούτο δεν μπορούσα να έρθω στην ώρα μου, να είμαι ακριβή και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η συνάδελφος ε, Κλάουδια Σμιτ, ε, από ό,τι άκουσα, δεν μπορεί να έρθει λόγω χιονιού στην Αυστρία και με παρακάλεσε να διαβάσω τη γνωμοδότησή τη. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση τη κοινή γεωργική πολιτικής μετά το 2020 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 έχει καταθέσει μια δέσμη νομοθετικών προτάσεων που αποτελείται από τρία συγκεκριμένα κείμενα και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται και στην επικεφαλίδα, αφορά στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση, ε, την άποψη δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το 2020. Η πρόταση Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα και μεταξύ άλλων ασχολείται και με τον ορισμό των οργανισμών που εμπλέκονται σε εθνικό επίπεδο. Ασχολείται με τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν όταν παραβιάζονται οι κανονισμοί. Ε, η άποψη τώρα της κυρίας Σμιτ. Σε γενικές γραμμές καλή η πρόταση της Κομισιόν, αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η άποψη της Επιτροπής Παρακολούθησης ε, να ε, υπάρχει καλύτερο έλεγχος της χρηματοδότηση. αυτό είναι μια καλή εξέλιξη και το σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, έχω επιφυλάξει όσον αφορά το ποιο αναλαμβάνει την ευθύνη του ελέγχου. Στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει αυτό τον έλεγχο όλο και περισσότερο στις εθνικές αρχές. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ε, μια κατανάγκη παραχώρηση μετά το 2020 στην κοινή γεωρική πολιτική ε, θα υπάρχουν αποδόσεις ε, μετά από περισσότερους ελέγχους και όχι γιατί γίνεται σεβαστό το νομικό πλαίσιο. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα αναλαμβάνει λιγότερες ευθύνες και θα εκπληρώνει λιγότερο τις υποχρώσεις. Εξελίξει όπως η Τσεχοσλοβακία κατέδειξαν ότι αυτό είναι λάθος δρόμος και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους. Εγώ λοιπόν για αυτό το λόγο κατέθεσα 15 τροπολογίες οι οποίες προβλέπουν από δίδεται περισσότερη ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν διατηρηθεί η πρόταση Επιτροπή ω έχει, αυτό θα σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν θα λαμβάνει πλέον στατιστικά δεδομένα ελέγχου από του οργανισμού πληρωμών των ε, κρατών μελών. Και αυτό σημαίνει ότι επίση θα μπορούσαν να ε, ακυρωθούν κάποιε πληρωμέ. Άλλε συνέπειε η Κομισιόν δεν θα μπορεί να ποσοτικοποιήσει σε ποιο βαθμό παραβιάζονται οι κανονισμοί. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι κάθετα αντίθετο με όλα αυτά που αναφέρονται στις συνθήκες, ότι σε τελική ανάλυση η Κομισιόν εκείνη η οποία έχει την τελική ευθύνη για τον προεπολογισμό. Εγώ με τις ε, τροπολογίες μου προσπαθώ να ε, επαναφέρω την ανάληψη ευθύνη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τροπολογίες μπορούν να κατεθούν μέχρι την Πέμπτη ε, στις 2 η ώρα. Τον Ιανουάριο θα ψηφίσουμε για την άποψη αυτή ε, δεν έχει ακόμα κατατεθεί και δεν έχει αποφασιστεί πότε θα συζητήθει το θέμα στην Γεωργική Επιτροπή, αλλά προβλέπεται μάλλον μέσα Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κάτμπαου. Κάτμπαχα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ έρχομαι από τα ανατολικά της Αυστρίας. Σε εμάς η κατάσταση δεν είναι τόσο κακή, άρα μπόρεσα να έρθω στην ώρα μου. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο κύριο Τσέλε για την παρουσίαση της άποψης της συναδέλφου κυρίας Σμιτ. Η κυρία Σμιτ και εγώ διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτή τη φορά μάλλον συμπίπτουν αρκετά οι απόψεις μας. Θεωρούμε ότι η πρόταση Επιτροπής οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής και νομίζω ότι οι προτάσεις που έχει κάνει και η κυρία Μούλερ από την Επιτροπή Γεωργίας είναι σωστές. Δηλαδή στο μέλλον ε, σε τελική ανάλυση η τελική ευθύνη θα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την άποψη της ε, κυρίας ε, Σμιτ. Εκ μέρου τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω την κυρία Μπόρχ Μαν, αλλά δεν ξέρω ποιο θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους. Σας ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένη. Νόμιζα ότι θα αφιερώνατε περισσότερο χρόνο στο, στα πρώτα σημεία της ημερήσια διάταξης. Σα ζητώ συγγνώμη λοιπόν για την καθυστερημένη αφήξή μου. Είδα πολύ γρήγορα τα όσα μας είπε ο κύριος Τσέλερα πριν από λίγο. Θα ήθελα καταρχά να σας πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τον οριζόντιο κανονισμό και το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρία Σμιτ. Προφανώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει ότι είστε υπέρ της επιχειρούμενη τροφής από ένα μοντέλο βασισμένο στη συμμόρφωση, ένα μοντέλο βασισμένο στις επιδόσεις. Πρέπει να σας πω ότι το νέο αυτό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται ουσιαστικά στον οριζόντιο κανονισμό και σχετική πρόταση, θέτει τις επιδόσεις ως ακρογωνίο λίθο για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Εστιάζουμε λοιπόν όλο και περισσότερο στι επιδόσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε το σύστημα αυτό κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ξεφύγουμε από το επίπεδο του μεμονωμένου δικαιούχου και να έχουμε καλύτερα μία ξεκάθαρη εικόνα των επιδόσεων σε επίπεδο κρατών μελών πλέον. Γι' αυτό το λόγο μέσω των επιδόσεων θα θέλουμε να δούμε πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νέου αυτού μοντέλου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής και από το σχέδιο γνωμοδότησης βλέπουμε βέβαια ότι έχουν ήδη προκύψει σε εσά κάποιες ανησυχίες. Θα θέλατε να επικεντρωθούμε περισσότερο στους μεμονωμένους δικαιούχους, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, τροποποίησεις από τις οποίες φαίνεται ότι εσείς έχετε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χάσει λίγο τον έλεγχο όσον αφορά τα μονομένα κράτη-μέλη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο οριζόντιος νέος αυτός κανονισμός παρέχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα μονομένα κράτη-μέλη και στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Συνεπώς λοιπόν θα έχουμε συστήματα διακυβέρνησης τα οποία θα συνεχίσουν να την χάνουν ελέγχου και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση. Επίσης, οι οργανισμοί διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη θα εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι. Θα χρειάζεται οι οργανισμοί αυτοί να δηλώνουν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν τηρούνται οι κανόνε και αν υπάρχει απαραίτητη συμμόρφωση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει με του ελέγχου που κάνει μέχρι τώρα. Θα έχουμε δηλαδή την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τι επιθεωρήσει και του ελέγχου. Όλοι οι έλεγχοι συμμόρφωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αφορούν όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Στο σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρεστε πολλές φορές σε ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και κυρίως τα οποία έχουν τονίσει διάφοροι δημοσιογράφοι, ερευνητές δημοσιογράφοι. Σας διαβεβαιώνουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να ελέγχει για το αν τα συστήματα λειτουργούν σωστά και αν δεν λειτουργούν σωστά θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπει το άρθρο 53. Όταν διαβάζουμε τώρα τις προτινόμενες τροπολογίες στο σχέδιο αυτογνωμοδότησης, ουσιαστικά μας ζητάτε να έχουμε ελέγχου συμμόρφωση σε επίπεδο δικαιούχων για κάθε ξεχωριστή ενίσχυση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα διτό σύστημα με επικαλύψεις, όπου θα πρέπει πέρα από το μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στη συμμόρφωση και το οποίο ζητάτε να επανεισάγουμε, να έχουμε και το μοντέλο βασισμένο σε επιδόσει, το οποίο εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώ αυτή την επικάλυψη θέλουμε να αποφύγουμε. Θεωρούμε ότι το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο μοντέλο το οποίο προτείνουμε για την κοινή γεωργική πολιτική ουσιαστικά βελτιώνει το σύστημα, διατηρώντα όμω τα ισχύοντα συστήματα ελέγχου. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Να αναφερθώ απλώς στην τροπολογία επαριθμών 6 για το άρθρο 46 όπου εδώ το σχέδιο γνωμοδότησης μας προτείνει το αποκομίζει να γίνει μπορεί να αποκομίσει, δηλαδή να έχουμε ένα may. Υπάρχει όμως στο κανονισμό ήδη ο όρος shall, λέγεται ότι για τους σκοπούς του άρθρου 127 του Δημοσιονομικού Κανονισμού η Επιτροπή μπορεί να αποκομίσει βεβαιότητα για την εξοπιστία τους από τις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης. Ουσιαστικά εδώ πέρα θέλουμε να βλέπουμε για ποιους ελέγχους που θα κάνουν οι οργανισμοί πιστοποίησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει εκθέσεις διασφάλισης της εξοπιστίας. Επίσης γίνεται μια αναφορά σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου στην ε, τροπολογία σας γίνεται μια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό το οποίο όμως ε, αποφασίστηκε στην ε, πρόσφατη απόφαση για τον κανονισμό Omnibus και που έχουμε στην πρόταση αυτή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα την χάνει ελέγχου από τα κράτη-μέλη, αλλά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη τις εκθέσεις που συντάσσει, που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εδώ ουσιαστικά απλώ ακολουθούμε τα όσα έχουν ήδη αποφασιστεί στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus. Είμαστε λοιπόν υπέρ, μάλλον χαιρόμαστε για το ότι είστε κι εσείς υπέρ για την στροφή αυτή που γίνεται από το μοντέλο που είναι βασισμένο στη συμμόρφωση προς ένα μοντέλο βασισμένο σε επιδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταφέρουμε να αποφύγουμε το δεύτερο αυτό επίπεδο επικάλυψη όσον αφορά το διοικητικό φόρτο, του διοικητικού ελέγχου, αφού είναι κάτι το οποίο ήθελε να πλουστεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προτινόμενη αυτή πρόταση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Η ξεκίνησε και βεβαίω ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσατε να μας καταδείξετε μία διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο. Ε, οι μεν λένε δεν έχετε δίκιο, οι άλλοι λένε δεν έχετε, δεν θέλουμε. Αυτό είναι το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε. Ε, το θέμα είναι ότι ακούσαμε καλές ιδέες, αλλά δεν ξέρω κύριε Μπόχμαν, θέλετε να ξαναλάβετε το λόγο. Ε, εγώ νομίζω ότι εδώ τίθεται και το θέμα της ε, αμοιβαίας ε, κατανόησης. Και θα ήθελα να εστιάσω στο γεγονός ότι τελικά ε, δεν καταργούνται τα συστήματα διαχείριση και ελέγχου στα κράτη-μέλη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βασικά λέμε ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα ίδια συστήματα όπω είναι αυτά ε, που ισχύουν σήμερα και θα συνεχίσουμε εμείς να ελέγχουμε ότι πράγματι όλα βαίνουν καλώς. Αλλά δεν θα φτάσουμε μέχρι και τον τελευταίο δικαιούχο. Εμείς θα διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν τα συστήματα και κατ' ουσίαν αυτό κάνουμε και σήμερα στους ελέγχους που διεξάγουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή δεν ελέγχουμε με μονομένους δικαιούχους, ελέγχουμε τα συστήματα, κατά πόσον λειτουργούν σωστά. Πάντως προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λύση όπου υπάρχει μία συνταγή για όλα και αν δει κανεί κάποιε κάποιες περιπτώσεις ε, αυτές, που αναφερθήκατε των ε, ερευνητών δημοσιογράφων, εκεί θα δείτε ότι οι κανόνε δεν γίνονται σεβαστοί γιατί δεν έχουν και πάντα νόημα κάτω από ορισμένε συνθήκες σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλο. Και η ιδέα είναι με αυτό το νέο μοντέλο περί απόδοσης, τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευελιξία για να μπορούν να διασφαλίσουν ότι πράγματι θα έχουμε καλή απόδοση, ε, θα έχουμε τα αποτελέσματα Λέγοντα που επιδιώκουμε και αυτό ε, θα το έχουμε προσαρμόσει σε ένα κράτος μέλος. Δεν θα έχουμε κάτι που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί όπως σας είπα με το τρέχον σύστημα υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κανόνες ε, δεν εφαρμόζονται και προβαίνουμε σε δημοσιονομικές διορθώσεις, αλλά κατ' ουσίαν αυτό βλάπτει την απόδοση. Και αυτό δημιουργεί και προκαλεί επικρίσεις κατά του συστήματος. Και η δική σας Επιτροπή και αυτή έχει καταθέσει μία έκθεση για το ε, διοικητικό άχθος ε, σχετικά με τους ελέγχους ε, και πρέπει να πω και εγώ, ναι, υπάρχει διοικητικό φόρτο, αλλά εμεί θέλουμε να πλουστεύσουμε του κανόνε και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι θα επιτυγχάνονται και τα ευκταία αποτελέσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι και θέμα κατανόησης, δηλαδή να γίνει κατανοητό ότι δεν απομακρυνόμεθα από ε, το ότι τα κράτη-μέλη τελικά θα έχουν τον έλεγχο και τη διαχείριση, ε, κάτι που κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στη γνωμοδότηση, ε, το υπονοεί η συγκήτρια. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να ζητήσουμε έναν, μία μέση οδό. Πρόεδρος, την εμπειρία την συλλέγει κανείς αν εξετάσεις συστήματα. Και τι διαπιστώνουμε, κάνουμε την εξής εμπειρία, ότι ε, κάποιες φορές ε, υπάρχει μια συστημική άποψη στα διαρθρωτικά ταμεία και πρέπει κανείς να απομακρυνθεί από αυτή. Και θέλω να επισημάνω ότι τα συστήματα ελέγχου ε, στα διαρθρωτικά ταμεία δεν αποκαλύπτουν πολλές φορές πολλά πράγματα. Και εμείς ανησυχούμε, φοβούμαστε ότι θα επαναληφθεί αυτό που το γνωρίζουμε ήδη από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπου δηλαδή καθαρά συστημικά είναι όλα τέλεια και αν δει κανεί μετά επιτόπου αυτή η έγκλη, αυτή η λάμψη θα μπώνει εξαφανίζεται. Αυτό μας ανησυχεί και μας ανησυχεί ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Και νομίζω τελικά αυτό προκύπτει από την όλη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα. Με δυσάρεστο τρόπο. Έχουν κατατεθεί πάρα πολλές ε, τροπολογίες και εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, Τέλο πάντων, ε, κρίνω ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Γνωρίζουμε επίσης ότι το θέμα με την κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι απλό και εγώ επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα αυτή η πολιτική δεν ήταν και τόσο κακή, ούτε και τόσο, σε τόσο δυσάρεστη θέση βρίσκονται οι γεωργοί. Αυτό το θέμα του να ε, χορηγούνται κονδύλια χωρίς κανένα έλεγχο, αυτό δεν θα υλοποιηθεί, δεν θα γίνει ποτέ. Θα δούμε λοιπόν ε, πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής θέλει το λόγο. Όχι, εγώ έχω την τυπική μου έκθεση και νομίζω και εκεί συζητιέται περίπου το ίδιο θέμα. Ωραία, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Ιανουαρίου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας πλέον, 10 ε, Ιανουαρίου μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ξανασυζητηθούμε το θέμα αυτό στις 28 και 29 Ιανουαρίου. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο σημείο υπερθυμών 6 της ημερήσιας διάταξης. Και είναι πάλι ένα θέμα για τη Γεωργία, τα στρατηγικά σχέδια. εσύ είναι ο ίδιο ο κύριος Τσέλερ αυτή τη στιγμή. Γνωμοδότηση δεν έχουμε λάβει ακόμα. Το λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Τσέλερ, ο συντάκτης της, μάλλον ο εισηγητής και συντάξει νομοδότηση. Ευχαριστώ. Η κοινή γεωργική πολιτική ξανά μας απασχολεί. Η δική μου γνωμοδότηση βέβαια τώρα αφορά τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κοινή γεωργική πολιτική. Κατά την άποψή μου είναι αρκετά επικριτική η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τα μελήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς αυτά υλοποιούνται. Είναι επικριτική, λέω, η έκθεση από πλευράς ελεκτικού συνεδρίου. Επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζει μεν το γεγονός ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να ενισχύσει ε, την ε, Ευρωπαϊκή Κοινή Γεωργική Πολιτική και να την προσανατολίσει καλύτερα στις επιδόσεις και σε κοινού στόχους αυτό το ακούσαμε και προηγουμένως στην γνωμοδότηση της κυρίας Σμιτ και το συζητήσαμε. Ήταν και δική μας άλλωστε επιθυμία και αίτημα από τις απαλλαγές των προπολογισμών των περασμένων ετών. Η κοινή γεωργική πολιτική να, φύγει, να ξεφύγει από μια μηχανή διανομής χρήματων και να περάσει σε ένα τομέα πολιτικής που ε, θα έχει περισσότερο κοινού πανευρωπαϊκούς στόχους και θα υπάγεται σε αυτούς και ακούγονται κυρίως περιβαλλοντικοί στόχοι που γράφονται στην έκθεση πώς υλοποιούνται αυτοί κατά αποδέμιση της κλιματικής αλλαγής και συνεισφορά της γεωργίας προς την κατεύθυνση αυτή. Πού καταλήγει όμως το λέει συνέδριο ότι δεν είναι αρκετές οι προτάσεις για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτών των επιδόσεων. Και η Επιτροπή Γεωργίας αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν πιο απλά κριτήρια, ε, απλουστευμένα κριτήρια για την κοινή πολιτική. Στραματική ενίσχυση ουσιαστικά να παίρνουν τα λεφτά με βάση την επιφάνεια και αυτά. Και μετά μας λένε αφήστε μας και στην ησυχία μας με όλα τα υπόλοιπα. Εμείς ε, τρέφουμε τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και αυτό θα πρέπει να σας αρκεί. Βέβαια, συμφωνούμε εμείς με το ελεκτικό συνέδριο να υπάρχουν σαφείς στόχοι μετρήσιμοι και συγκεκριμένοι και οι φυστάμενοι στόχοι να αξιολογηθούν και να συνδεθούν ε, με τις επιπτώσεις ε, και ε, τα αποτελέσματα. Να μην έχουμε δηλαδή μόνο μια τσέπη από την οποία να βγάζουμε χρήματα, να υπάρχει και ένα input, δηλαδή να, να μαθαίνουμε τι γίνονται αυτά και ποιες είναι οι επιδόσεις και να ελέγχεται κατά πόσο οι στόχοι τους οποίους ε, θέτουμε και ε, σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς θα έχουν υλοποιηθεί. Ε, δηλαδή, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες, περισσότερα κίνητρα για επιδόσεις. Έχω κάνει και τροπολογίες με στόχο να έχουμε δεσμευτική συμπερίληψη ε, και λήψη υπόψη των όσων λέει το ελεκτικό συνέδριο σε μια μελλοντική γεωργική ε, πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς δείκτες που να μετρούν και να αξιολογούν τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και η κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο λίγο πιο διαφανή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν στοιχεία αξιόπιστα και ε, συγκρίσιμα, ας πούμε, ως προς το εισόδημα και το, το υπολογισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Γιατί μέχρι τώρα αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί και ήταν και πάντα πρόβλημα στις διαδικασίες ε, χορήγησης απαλλαγής. Επίσης, η ποιότητα και ο τρόπος λειτουργίας, καθώς επίσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γεωρικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να μας απασχολήσει λίγο πιο στενά. Είναι ακόμα η παραδοσιακή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση ε, που δημιουργεί απασχόληση, φροντίζει το τοπίο και την ύπεθρο εκεί στις περιφέρειες ή μήπως εδώ και καιρό όλα αυτά έχουν γίνει μεγάλες βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις ε, που τελικά ανήκουν και σε ε, ανώνυμες επενδυτικές εταιρείες. Και η γεωργική πολιτική δεν είναι απλώς μια υπόθεση επιδοτήσεων, αλλά μπορεί κανείς να βγάλει και καλά λεφτά. Άρα τίφτει γενικά το θέμα των επιδοτήσεων, είναι σκόπιμες αυτές. Χρειάζεται λοιπόν πιο αποτελεσματική γεωργική πολιτική και για να γίνει αυτό διαφανή κριτήρια, ε, ποιότητα, σχέδια στρατηγικής για να κρίνουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Σε αυτό καταλήγει το ελεκτικό συνέδριο και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάντεμπαχ. Τώρα είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μια γνωμοδότηση που δεν την έχουμε στα χέρια μας και να τοποθετηθούμε. Πάντως, γενική συζήτηση καλό είναι να κάνουμε για να δούμε πώς αξιολογείται γενικά η κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει εδώ ένα σημείο ε, που θέλω να θέσω ε, σε σχέση με τόσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δεχόμαστε εμεί αυτή την κατηγορία. Το κατηγορείται το Κοινοβούλιο ότι θέλουμε μία λύση για όλου. Όχι, είδαμε στο παρελθόν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ε, σκόπιμο. Και δεν ήταν μόνο η κριτική του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και των βουλευτών πάγια. Το πρόβλημα ποιο είναι. Αν έχουμε μια κοινή, και ο τόνος είναι στην κοινή ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, θα πρέπει αυτό να το δούμε ως ένα εργαλείο καθοδήγηση και η καθοδήγηση θα πρέπει να είναι κοινή. Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό κατά τη γνώμη μου επικρίνει το ελεκτικό συνέδριο. Ότι στι προτάσει γενικώ και απλώ με το μανδύα και πρόσχημα της επικουρικότητας αφήνουμε να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο τα κονδύλια ώστε να μην μπορεί πια να τα ελέγχει ούτε το ελεκτικό συνέδριο ούτε το κοινοβούλιο, γιατί είναι πολύ λίγα τα ε, συγκεκριμένα μετρήσιμα κοινά κριτήρια και είναι πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Το κάθε κράτος μέλος δηλαδή, ακόμα περισσότερο σε ε, χώρες με ομοσπονδιακή δομή που έχουν ομόσπονδα κρατήδια ή όπως αλλιώ λέγονται οι περιφέρειες ή ενότητες. Δεν έχουμε ενιαία αντιμετώπιση. Και εκεί συμφωνούμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστώσεις από εκεί και πέρα με βάση ποια κριτήρια ε, γίνεται αξιολόγηση. Και πού είναι και το επιστημονικό υπόβαθρο ε, όταν έχουμε ένα σύστημα τόσο κατακαιρματισμένο και τόσο διαφοροποιημένο. Αυτό που λέμε τώρα μπορεί να... Ε, ε, μάλλον αυτό που μας παρουσιάσατε μπορεί να ενδείκνεται για το απότερο παρελθόν, αλλά, μέλλον, αλλά όχι για τη σημερινή περίοδο και την επόμενη περίοδο. θέλουμε αξιοπιστία και συγκρισιμότητα σε πολύ σύντομο χρόνο. Και εκεί είναι το πρόβλημα και ο κίνδυνο. Στόχο, δεν είναι να έχουμε μία λύση για όλους, αλλά μια κοινή κατεύθυνση της κοινή γεωργική πολιτικής και να μπορούμε αυτά να τα μετρούμε και να τα ελέγχουμε και βεβαίω να προσανατολίζονται στα αποτελέσματα, αλλά για αυτό το σκοπό ακόμα μας λείπουν οι δείκτες. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Σίφλα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα ε, και να αναφερθώ και σε αυτά που είπε η παρακαθήμενή μου. Κοιτάξτε, για μας ε, τρία είναι τα βασικά θέματα που μας καθοδήγησαν. Το πρώτο, οι μακροχρόνιες όλες αυτές οι συζητήσεις για την απλούστευση του συστήματος. Αυτές όμως οι συζητήσεις δεν οδήγησαν πουθενά. Και ως εκ τούτου συμπεράναμε ότι αν ε, πραγματικά θέλουμε ουσιαστικές απλουστεύσεις, τότε θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα, σε ένα σύστημα που θα είναι προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα να μετράει για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία ορίζουμε με σαφήνεια θα τα ελέγχουμε, αλλά να μην ορίζουμε και την τελευταία λεπτομέρεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεγαλύτερη επικουρικότητα, μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών στην τελική διαμόρφωση, βέβαια με βάση κοινού στόχους και κοινέ αρχές. Το δεύτερο, όσον αφορά τους κοινού στόχους, έχουμε ε, τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής που τους ορίζουμε με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, από ό,τι ήσχε μέχρι τώρα, ε, για να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα ε, του γεωργικού χώρου. Και καθορίσαμε και κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Είτε είναι το κάπινγκ, είτε η αιρεσιμότητα, είτε οι αρχές για τη διαχείριση κινδύνων. Αυτά λοιπόν είναι καθοριστική σημασία θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τρίτη βασική αρχή. Κατά την εφαρμογή θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, συγκεκριμένο περιθώριο όπου οι στρατηγικοί στόχοι της κοινή γεωργική πολιτική βεβαίω και θα πρέπει να προσανατολίζονται στους νέους στόχους, αλλά παράλληλα και να εστιάζονται σε μια ενδελεχή ανάλυση και έλεγχο του τι πρέπει να γίνει επίτόπου. τόπου. Και εκεί παρισφρεί το διαφοροποιητικό στοιχείο. Όσον αφορά στην εφαρμογή των στρατηγικών προγραμμάτων της ε, ΚΑΠ, πράγματι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, να γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος όσων έχουν επιτευχθεί και γι' αυτό προβλέπουμε τους ετήσιους ελέγχους, οι οποίοι σε τελική ανάλυση διασφαλίζουν ότι θα έχουμε δείκτες που αφενός θα είναι διαχειρίσιμοι, αφετέρου όμως και οι δείκτες αυτοί θα είναι καταλητική για το τι γίνεται τελικά με τους στόχους. Με αυτούς λοιπόν τους δείκτες ε, στα κράτη-μέλη ορίζονται ε, ορόσημα και ορίζονται και θέματα που μπορούν να βοηθήσουν για να υπάρξει πρόοδος. Υπάρχει και το εξή ε, υπάρχει μια καινοτομία, ότι κατά την εφαρμογή κατά την εφαρμογή ε, και του συστήματος ε, που προβλέπεται στην εφαρμογή θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά έγκαιρα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προγράμματα δράσης όπου ε, ορίζονται τα ορόσημα που σας είπα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια απόκληση από το στρατηγικό πρόγραμμα. Διαφοροποίηση λοιπόν που συμβαδίζει με τη μεγαλύτερη επικουρικότητα, κοινέ αρχές, κοινή στόχοι που διασφαλίζουν το κοινό στοιχείο της πολιτικής και σαφής ε, επιδίωξη των στρατηγικών πάνω σε αιτήσια βάση για να διασφαλίζεται και πάλι ότι ο προσανατολισμός και η διαφοροποίηση πράγματι εφαρμόζονται ως έχει προβλεφθεί. Και αυτό μπορεί ή μάλλον πρέπει να υπάρχει σε έναν αιτήσιο έλεγχο. Όσον αφορά τώρα τους δείκτες και τα αποτελέσματα τα οποία ε, καλύπτουμε μέσα από τους δείκτες, ε, θα πρέπει όλα αυτά να είναι διαχειρίσιμα. Και ο έλεγχος ε, θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην διαχείριση. Γιατί τι να το κάνουμε αν σε αιτήσια βάση εξετάζουμε την βιοπικιλότητα όπου ξέρουμε ότι από την παρέμβαση μέχρι το τελικό αποτέλεσμα ε, προκύπτει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Ή ε, στα μέτρα προστασίας των υδάτων, τα νητρικά άλατα. Αυτά χρειάζονται χρόνια για να ε, φανούν τα αποτελέσματα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίζονται τα επιστημονικά κριτήρια. Και αν κατά την εφαρμογή διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει πρόοδος, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δημιουργείται αυτό το αδιέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση αυτή να ε, συντονιζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να λύνουμε τα προβλήματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να σα πω, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι προτάσει τη Επιτροπής, το γιατί κάνατε αυτέ τι προτάσει. Μόνο που ξέρετε, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σα. Ε, δηλαδή ότι με τι προτάσει που καταθέσετε θα επιτύχετε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Γιατί, διότι μέχρι τώρα το πρόβλημα είναι το ότι στον γεωργικό τομέα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και πολλέ διαφορέ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτές λοιπόν οι διαφορές οδηγούν στο ότι ορισμένα κράτη-μέλη τελικά εφαρμόζουν τη γεωργική τους πολιτική εις βάρος ενός άλλου κράτους μέλους. Ε, αυτό πρέπει να το δούμε. Να δούμε το πόσο πολύ θέτει σε κίνδυνο αυτή η κατάσταση την συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοώ ότι η κλίμακα το μέγεθο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ α πούμε στην Πάρη Βιτεβέργη όμω ε, ξέρω ότι θέλουμε να ε, βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, όμω οι μεγάλε επιχειρήσει τελικά τι καταπιέζουν, τι πιέζουν και αυτό ε, στο μέλλον θα επιταθεί περισσότερο. Δηλαδή αν το μέγεθο ή κλίμακα παίζει ρόλο, φοβάμαι ότι αυτό θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Μιλήσατε για το κάπινγκ. Εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξη όσον αφορά το θέμα αυτό. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι τι ακριβώς γίνεται ε, για να δούμε πώς ακριβώς επιμερίζονται τα κονδύλια. Ε, πρέπει να σας πω ότι είχα λόγο βέβαια, ασχολήθηκα σε βάθος ε, με την Τσεχοστροβαχία. Βέβαια η αεροπορική εταιρεία με εγκατέλειψε στο αεροδρόμιο. Η και αν ε, καταλήξουμε και πούμε ότι τελικά παίρνουμε μόνο το 70% των κονδυλίων, νομίζω ότι δεν επιτυγχάνουμε τίποτα. Γιατί ε, έχουμε την Τσεχία, την Τσεχοσλοβακία, έχουμε Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία, οι οποίες ε, έχουν τελείως διαφορετικές δομές και θέλω να ρωτήσω στις προτάσεις εσεί ως Επιτροπή τι δυνατότητες βλέπετε. Επειδή βλέπω ότι κανείς άλλο δεν θέλει το λόγο θα ήθελα να σα ξαναδώσω το λόγο πριν όμως θα λάβει το λόγο στην άλλη κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, και στη δική μας τη χώρα, στη Γερμανία, έχουμε διαφορά, διαφοροποίηση στις δομές και αυτά που είπατε κυρία Πρόεδρε για κάποια κράτη, αυτά είναι κράτη τα οποία έχουν πίσω τους ε, σοσιαλιστική γεωργία. Ήταν μεγάλα, τεράστια κολχόζ. Στην Ανατολική Γερμανία μάλιστα καταβλήθηκε προσπάθεια ε, να δημιουργηθούν κατά δεκαετία του 70 συνεταιρισμοί όπου πολλά χωριά συνενώθηκαν και είχαν μία και μόνο επιχείρηση. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση στις περισσότερες ε, περιπτώσεις, το 91-92 παρότι άλλαξαν οι πολιτικές συνθήκες, δεν άλλαξε η πραγματική κατάσταση. Τώρα υπάρχουν οι ίδιες μορφές, ονομάζονται ανώνυμες εταιρείε, έχουν πάρει κάποια μορφή στα πλαίσια του αστικού δικαίου, αλλά κατ' ουσίαν το μέγεθος, η κλίμακα έχει παραμείνει. Εσεί αναφερθήκατε στη Βάδεντεμπέργη. Εγώ θα μιλήσω για τον Παρδιμπούργο ή για τη Σαξονία Άνχαλτ. Εκεί έχουμε μικρού ε, γεωργού οι οποίοι προσπαθούν να συστήσουν γεωργικές επιχειρήσεις, τοπικές, αλλά ε, εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες δυσκολίες γιατί σε τελική ανάλυση στα ε, κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας γι' να το λόγο ακριβώς υπάρχουν και δύο γεωργικές ενώσεις αυτά τα οποία περιγράψετε σε σχέση με τον επιμερισμό, αυτή είναι η τρέχουσα πολιτική. Δεν πρέπει να το κρύβουμε. Ε, σε αυτή την πολιτική ε, υπάρχει αυτό το θέμα που όλοι μας ε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Με τις εξή συνέπειες, ότι στην μελλοντική γεωργική πολιτική, όπως και εσείς είπατε, για αυτή τη μελλοντική γεωργική πολιτική, τους κοινού στόχους τους βάζουμε πρώτους και αυτά που θέλει να επιτύχει το στρατηγικό σχέδιο, αυτό πρέπει να αιτιολογείται με τους στόχους. Δεν ισχύει μόνο για το δεύτερο πυλώνα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά για το σύνολο της γεωργικής πολιτικής. Ως εκ τούτου έχουμε και κάποια συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Έχουμε την ενίσχυση των νέων γεωργών. Έχουμε τις συνεργασίες μέσα από τα οικολογικά προγράμματα. Όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν ε, αιτιολογούμενα όμως, τεκμηριωμένα περισσότερο θα έλεγα και ε, νομίζω ότι με αυτή την προσέγγιση είμαστε πολύ πιο κοντά στη σωστή πολιτική. Προτείνουμε βέβαια και το κάπινγκ, το οποίο σε τελική ανάλυση και αυτό οδηγεί σε σωστή κατεύθυνση το θέμα του επιμερισμού των κονδυλίων. Βεβαίω ε, δεν θα ανατρέψουμε τα πάντα, το σύστημα που υπάρχει μέχρι τώρα, απλά θέλουμε να υπάρχει μία ε, πιο σωστή κατεύθυνση που να βασίζεται σε τεκμηρίωση. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα που απαντήσατε, αλλά στο πρώτο δεν απαντήσατε. Που το ξέχασα κι εγώ. Κι εγώ το ξέχασα, λέει η πρόεδρος α, ε, τον ανταγωνισμό των κρατών μελών ανάμεσά τους λόγω της διαμόρφωσης της ε, γεωργικής πολιτικής. Εδώ έχουμε ένα ε, σαφές πλαίσιο κοινών στόχων και υπάρχει η εξή προϋπόθεση. Οι τα στρατηγικά σχέδια της ΓΑΠ βεβαίως και πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια τοπική προσέγγιση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να αιτιολογούν το πώς θα επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε έχουμε μια σαφή προϋπόθεση η οποία θα οδηγήσει σε συνοχή ανάμεσα στα κρατη Υπάρχει και η αιρεσιμότητα σε σχέση με το περιβάλλον, η οποία θέτει ελάχιστες κοινέ προδιαγραφές. Και έχουμε και μία διαδικασία όπου με την ε, υιοθέτηση των προγραμμάτων της κοινή γεωργικής πολιτικής, όπως ακριβώς το γνωρίζουμε από το δεύτερο πυλώνα, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να διορθώσουμε, να συγκρίνουμε, γιατί γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν θέματα όπου πράγματι μέσα από ένα μηχανισμό συνένεσης και συνοχής επιτύχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιτύχαμε δηλαδή κάποια συνέπεια, κάποια συνοχή ε, στο αποτέλεσμα και αυτό οφείλεται στο ότι εγκρίθηκαν μέτρα τα οποία οδηγούν περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση της συνοχής. Βεβαίως υπάρχει και η εξή αρχή. Η συμπληρωματικότητα πρώτος δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να αιτιολογείται από τον στρατηγικό προγραμματισμό με τους νέους στόχους και γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα, όπου ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας αντιμετωπίζονται δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και όπου ε, στον πρώτο πυλώνα δεν υπάρχουν καν ίση ώρα ανταγωνισμού, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε. Ωραία, λοιπόν. ευχαριστώ. Για να δούμε τι θα προκύψει. Δεν το λέω καθόλου ηρωνικά και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Κυριολεκτό, γιατί είναι σημαντικό για μας. Αν κοιτάξω τι γίνεται στις διοικήσεις, στη Γεωργία, σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει μεγάλη διασύνδεση μεταξύ Γεωργίας και διοίκησης. Έχω πεμπολίσει εδώ και καιρό το όνειρο ε, να ελέγχει η διοίκηση τη γεωργία. Έχει παγιωθεί αυτή η διασύνδεση και υπάρχει και μια περαιτέρω δυσκολία στη διαχείριση και στη διαδικασία για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων. Και αυτή θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ουδέτερο αξιολογικά. Και υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν βλέπονται. Δεν ξέρω, ε, έχετε προβλέψει τίποτα για αυτή την επιπλέον δυσκολία. Ναι, όντως, στο κείμενο το νομοθετικό έχουμε σαφείς κανόνες για την εταιρική σχέση και τη διαφάνεια στην προετοιμασία ε, όσο και την εκτέλεση των στρατηγικών προγραμμάτων θα συμμετέχουν και τα συναφή γειτονικά υπουργεία όπως είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι ενώσεις και οι σύνδεσμοι. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να υπηρετήσει τη διαφάνεια και την ανοιχτή διαδικασία. Μάλιστα. Ε, τελειώνει εδώ η συζήτηση, αλλά συνεχίζεται η ιστορία, θα μας απασχολήσει. Δεν θέλω να κάνω τροπολογίε που να καταστρέψουν το σύστημα για να δούμε να αρθροποδήσει και πώ θα λειτουργήσει και τι θα γίνει ε, στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Και εδώ έχουμε μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών που είναι η 10η Ιανουαρίου. Κυρία Τσέλερ, την γνωμοδότηση πότε θα τη δούμε. Βεβαίω θα πάρετε και το λόγο για να κλείσετε ω συντάκτη γνωμοδότηση. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, είναι σωστή η κατεύθυνση το μήνυμα το ακούμε, ναι, αλλά γνωρίζουμε και τι φρονούν οι συνάδελφοί μας στην Επιτροπή Γεωργίας. Θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου κάποια στιγμή. Και όπως σας είπα για τις τροπολογίες, έχω κάνει ε, τροπολογίες για τη, στη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου. Τις επόμενες ημέρες θα πάρετε και τη γνωμοδότηση. Έχει γίνει προεργασία από εμά, αλλά από την Επιτροπή Γεωργίας Σιγή Ιχθείος. Δεν ξέρω τι κάνει η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή και τι σκέφτεται, τι κατεύθυνση θέλει να δώσει σε αυτή την υπόθεση. Είναι σημαντικό όμως, διότι θα πρέπει σήμερα να πάρουμε τη γνωμοδότηση, γιατί 10 του μηνός λίγη προθεσμία και δεν έχουμε καν έκθεση. Ε, για να, πώς θα κάνουμε τροπολογίες. Πρέπει να μας δώσετε τη γνωμοδότηση αν γίνεται και σήμερα για να προλάβουμε. Ωραία. Ε, πάμε στο σημείο 7 τώρα. Ε, στην ε, συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου με τον Επίτροπο κύριο Οίτιγκερ, καλωσορίσαμε τον κύριο Κραφ, τον εσωτερικό ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε έπρεπε να, να συζητήσουμε τη δική του έκθεση. Αυτό αναβλήθηκε λόγω της συνάντησης με τον κύριο Ιούτιγκερ. το 2018, 661 λέγεται το έγγραφο εργασία και 421 ε, 429, συγγνώμη, τελικό. Είναι σημαντικές οι προφορίες που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και ευχαριστώ που ήρθατε ξανά στην Επιτροπή. Αλλάξτε, βλέπω γυαλιά. Με γεια και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Δεν ξέρω, θέλετε να μας παρουσιάσετε σύντομα την έκθεση, γιατί δεν είχατε καν την ευκαιρία μέχρι τώρα. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη δική μου, από τη δική μου πλευρά σας εύχομαι ότι καλύτερο για ένα επιτυχές 2019 ε, και σε εσά και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, εξαιτία της ακρόση του Επιτρόπου Έτιγκερ πριν από τη δική μου την παρέμβαση Είχαμε ελάχιστο χρόνο για να καταφέρουμε να υπησέλθουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε για την έκθεσή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα για να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο για το 2017. Όπω ξέρετε, σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια τη διαδικασία απαλλαγή υποβάλλει μια ετήσια εκθέση όσον αφορά τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετικέ συστάσει και δράσει που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και είπατε πολύ σωστά ότι δεν υπήρξε η δυνατότητα να κάνουμε μια αρχική παρουσίαση των συστάσεων αυτών και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση αυτή καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι δεσμεύεται για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία γιατί η έκθεση δείχνει με έναν ιδιαίτερα ανοιχτό και διαφανή τρόπο τα συστήματα τα οποία εφίστανται, καθώς επίσης και τα θετικά στοιχεία τους αλλά και τις αδυναμίες τους. Η έκθεση επίσης αυτή καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφασιστική δράση προκειμένου να θεραπεύσει τα δύναμα σημεία των συστημάτων αυτών εσωτερικού ελέγχου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας δίνουμε περισσότερες πληροφορίες στο πρώτο τμήμα του Αγγράφου Εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο, όπω ξέρετε, συνοδεύει την επίσημη έκθεση εσωτερικού λογιστικού ελέγχου σε ένα συγκεκριμένο κοιτίο, πίνακα μάλλον, βλέπετε τη συγκεκριμένη δράση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου που ολοκληρώθηκε το 2017. Καθότι εγώ είμαι ο εσωτερικός ελεγκτής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017, αφού ήταν η πρώτη έκθεση που υπέβαλα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνανε υπό τη δική μου την ευθύνη. Συνεπώς λοιπόν θα ήθελα να σε εξηγήσω λίγο περισσότερο πώς εφάρμοσα τις απαιτήσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων που θα πρέπει να εφαρμόζονται και στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ξέρετε ότι εδώ πέρα δεν είχαμε εμπλοκή άλλων φορέων όσον αφορά την έκθεση αυτή εσωτερικού λογιστικού ελέγχου που χρειάστηκε να γίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γιάλα Σέντερ που ήταν ε, η συγγήτρια για την απαλλαγή του 2017 ήδη στις 27 Σεπτεμβρίου μου έθεσε κάποια ερωτήματα όσον αφορά το ζήτημα αυτό και τις απάντησα τότε. Καθότι όμως οι ε, απαιτήσει που προκύπτουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Θεωρώ ότι θα πρέπει εκ νέου να σα παρουσιάσω σφαιρικά τα μέτρα τα οποία ανέλαβα. Βάσει λοιπόν των ε, οδηγιών που ε, εξέδωσα στις 7 Μαρτίου 2017, η εποπτεία του ελέγχου αυτού ήταν στα χέρια του κύριου Ντράφα Μέισον, ο οποίο ήταν ο πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και νυν επικεφαλής του IFBS, του νέου οργανισμού δηλαδή για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Επίσης, η Επιτροπή ABC ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις που κάνουμε και την εφαρμογή των συστάσεων αυτών. Στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής ε, συνεδρίασης της APC στις 6 Απριλίου αλλά και στις 3 Μαΐου του 2017 ελήφθησαν οι συστάσεις αυτές υπόψη. Η Επιτροπή επίση έλαβε υπόψη της την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται για το 2017 στην πρώτη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2017 καθώς επίσης και συνεδρίαση που έγινε το Μάιο του 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δράσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και είπε η Επιτροπή επίση ότι τα κατάλληλα μέτρα ελήφθησαν προκειμένου να υπάρχει ανεξαρτησία, ε, νομιμότητα για τους ελέγχους που ε, έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε στο παράρτημα επαριθμών 6. Πρωτού σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα πορίσματα των συγκεκριμένων αυτών εσωτερικών ελέγχων, θα ήθελα να κάνω πρώτα μια σφαιρική παρουσίαση του ε, ελέγχου του 2017. Μέχρι τις μέχρι το τέλος την 31η Ιανουαρίου του 2018 ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συστάσεων είχε εφαρμοστεί. 148 ήταν οι έλεγχοι τα καθήκοντα, τα 54 ήταν έλεγχοι, τα 19 ήταν συνέχεια και παρακολούθηση των δράσεων και των συστάσεων, δύο ήταν αναθεωρήσεις και δύο ήταν παροχή συμβουλών. Το 2017 η ΆΙΕΣ έκανε 199 συστάσεις. Οι 107 γίνανε απόλυτα δεκτές και οι δύο εν μέρη δεκτές. Όλοι οι ελεγχόμενοι υπέβαλαν σχέδια δράσης τα οποία υποβλήθησαν εν συνεχεία και εξετάστηκαν από την EIS. Εν γέννη απαιτείται χρόνος προκειμένου να εφαρμοστούν τα σχέδια δράσης. Επομένω, δεν θα ήταν λογικό να επικεντρωθούμε τόσο στην εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης για το 2017. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω περισσότερο τη συνέχεια που δόθηκε στις 1034 συστάσεις από το 2013 στο 2017. Από τις συστάσεις αυτές, οι 1.476 εφαρμόστηκαν, ένα 80% δηλαδή των συστάσεων, οι 359 είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 20%, ενώ 121 συστάσεις εκκρεμούν ακόμα και έχουμε και 12 πολύ σημαντικές συστάσεις 0,7% δηλαδή, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε δηλαδή μια καθυστέρηση πάνω από 6 μήνες σε σχέση με την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής. Η IS προχώρησε σε παρακολούθηση 136 από τις 147 συστάσεις, δηλαδή είναι 92%. 95% έκλεισαν από την EIS και ένα 5 μόνο της 100 των συστάσεων αυτών παραμένουν ανοιχτές. Στο δεύτερο τμήμα του Γράφου εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε λεπτομερεί πληροφορίε όσον αφορά την συνέχεια που έδωσε σε συστάσει η EIS. Θεωρεί εν γέννη ο οργανισμό αυτό ότι η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων είναι ικανοποιητική και μπορεί να συγκριθεί ικανοποιητικά με τα προηγούμενα έτη. Θα πρέπει όμω να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στι ε, κρεμεί συστάσει που ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί και για αυτέ περισσότερε πληροφορίε μπορείτε να βρείτε στο υπαριθμό 3 ε, τμήμα του εγγράφου εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να περάσω τώρα στα συμπεράσματα με βάση τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο του 2017, όπω έγινε από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Να επικεντρωθούμε δηλαδή στο έτο 2017 οι συστάσεις του AES όσον αφορά τις επιδόσεις θα μας απασχολήσουν σε ένα πρώτο επίπεδο και έπειτα οι συστάσεις όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική διαχείριση. Όσον αφορά το πρώτο βασικό τμήμα, της, τον έλεγχο δηλαδή των επιδόσεων, ως προς αυτό και εγώ αλλά και οι υπόλοιπε ομάδες ελέγχου βοηθήσαμε τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντοπίσουν συγκεκριμένου τομεί περαιτέρω βελτίωση. Το 2017 επικεντρωθήκαμε σε σημαντικά ζητήματα όπω ζητήματα διακυβέρνηση, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ζητήματα ασφάλεια του τομέα πληροφορική, καθώ επίση και οι ε, τομείς εκείνης στους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει άμεση έμεση ή συντρέχουσα αρμοδιότητα, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις συγκεκριμένων τομέων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπετε στα συμπεράσματα ότι σε πολλού τομεί υπάρχει περιθώριο βελτίωση, αλλά ότι σε πάρα πολλού τομεί έχουμε ήδη κάποιε πολύ ισχυρέ δομέ. Όταν προκύπτουν ζητήματα, τότε προβλέπεται κάθε φορά ένα σχέδιο δράση προκειμένου να θεραπεύσουμε και να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Η ΑΕΣ είναι ικανοποιημένη με τα συμπεράσματα αυτά. Στο πρώτο τμήμα του εγγράφου εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να δείτε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτά τα σχέδια δράση. Όσον αφορά τη δεύτερη σημαντική πτυχή, που είναι η χρηματοοικονομική διαχείριση και η διαχείριση των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν γέννη. Ως προς αυτό υπάρχει μια γενικότερη γνωμοδότηση για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με τη συμμόρφωση των γενικών ελέγχων τη και που λαμβάνει υπόψη και άλλες πηγές. Όπως γνωρίζετε, ο εξωτερικός μας ελεγκτής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και ο εσωτερικός ελεγκτής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν προβεί για το 2018 σε μία πανομοιότυπη γνωμοδότηση. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι λειτουργούν τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι τομεί στου οποίου εντοπίζονται ακόμα αδυναμίε. Ω εσωτερικό λογιστικό ελεγκτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέδωσα μια θετική γνωμοδότηση, αιτιολογημένη όμω υπάρχουν συγκεκριμένε επιφυλάξει όσον αφορά το, τις και τα προγράμματα εργασία τα οποία υποβάλλουν οι γενικοί διευθυντέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έλαβα υπόψη μου επίση τους εκρεμείς κινδύνους, καθώς επίσης και τις διορθώσεις που γίνονται σε επίπεδο ετήσιων προπολογισμών. Και γενικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι προπολογισμοί της Ευρωπαϊκής επιτροπή είναι αρκετά έγκυροι και ορθοί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση, σαφώ υπάρχει, αλλά εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι τα συστήματά μα είναι ορθά και αποδοτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει προβλήματα και θεραπεύει τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να θίξουμε, το οποίο το εντόπισε και στην έκθεσή μου για το προηγούμενο έτος, το ότι θα πρέπει να δοθεί πιο μεγαλύτερη έμφαση, ιδίω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ελέγχει, να λαμβάνει υπόψη τη διάφορου διαμεσολαβητέ, όπω για παράδειγμα τρίτε χώρε οι άλλοι τρίτοι οργανισμοί εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα και η συνδρομή των ανεξάρτητον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορούν να ελέγχουν τη διαμεσολάβηση αυτή και να δίνουν την απαραίτητη καθοδήγηση οι γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική επιτήρηση, εποπτεία, μια δραστηριότητα παρακολούθησης προκειμένου αυτές οι, ε, αυτοί οι εξοδοτημένοι εξωτερικοί φορείς όντως εφαρμόζουν ικανοποιητικά τα προγράμματα στην πράξη και ότι όντως προασπίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες που έλαβα από διάφορους εξωτερικούς φορείς καταδεικνύουν ότι όντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την επιτήρηση των οργανισμών αυτών. Στα συμπεράσματα επίσης του ελέγχου που έγινε από τον Διεθνή Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές συμβουλές οι οποίες πηγαίνουν ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι έχουμε έξι επιτρόπους και τρεις εξωτερικούς εκπροσώπους. Υπό την προεδρία του κυρίου Τίμερμανς, η ΑΕΣ έδωσε και θα συνεχίζει να δίνει πολύ σημαντική προσοχή στην ποιότητα των λογιστικών ελέγχων, καθώς επίσης και στην έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεών της από τις Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πορίσματα των ελέγχων αυτών να λαμβάνονται εγκαίρως υπόψη και επίσης οι γενικές διευθύνσεις να προβαίνουν σε συγκεκριμένες διορθωτικές πράξεις. Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μου αυτή, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι τόσο η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, αλλά και η Αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανεξελίξη Έλεγχο, προσπαθούν κάθε φορά να εντοπίζουν τις αδυναμίες και με έναν αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο να προβλέπουν συγκεκριμένες διορθωτικές πράξεις. Οι Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε φορά που αντιμετωπίζουν αδυναμίες, που εντοπίζουν μάλλον αδυναμίες σε οποιοδήποτε τομέα, αναλαμβάνουν την δέουσα διορθωτική τι δέουσε διορθωτικέ πράξει. Λαμβάνουμε υπόψη επίση και τι προηγούμενε συστάσει που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και είμαι πεπισμένο ότι με βάση τα συμπεράσματα τη έκθεση του 2017, καθώ επίση και μέσω των συστάσεων τη Επιτροπή τη CIS, τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προφανώς είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι έχουμε μια πολύ καλή εντύπωση και καλή εικόνα ότι όταν ανακύπτουν προβλήματα λύνονται κιόλα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, συμφωνούμε μαζί σας και σας ευγνωμονούμε που μας το λέτε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μερικά σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να τα συζητήσουμε. Η κυρία Ινέσα Γιάλα έχει το λόγο, η συγκήτρια για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους που έρχεται με μεγάλες προκλήσεις και πολλές και ελπίζω όλοι να είμαστε υγιείς και να έχουμε ενέργεια να τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ τον κύριο Κραφ για την πρώτη ε, δική του έκθεση, θα τη χαρακτηρίζα έτσι, η ίδια του έκθεση. Είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία ε, για ε, την απαλλαγή για το 2017 για την έκθεσή μου. Καρπός λοιπόν αυτής της εργασίας και των όσων μόλις μας είπατε είναι το εξής. Βέβαια αναγνωρίζω πάντα ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και έχουμε αναγνωρίσει τη δουλειά που έχει γίνει δεν χειροτερεύουν τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, μετά από τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το λέμε στους πολίτες ότι υπάρχουν και θετικά και θα πρέπει να τα αξιολογούμε, να τα τονίζουμε, να τα επενούμε και να προχωρούμε. Και όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο ξέρουμε τι απομένει να γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία προβληματάκια. Το πρώτο είναι αυτό στο οποίο και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε Εγώ το... Ε, έχω δει ε, αυτό που λέγεται ε, έμεση διαχείριση. Είδαμε τη συνυπευθυνότητα, τη συνδιαχείριση με τα διαρθρωτικά ταμεία και πώς γίνεται με τα κράτη-μέλη και πώς πρόβλημα υπήρχε για να τα συντονίσουμε, να τα ε, βελτιώσουμε και με την αποκέντρωση και με την άμεση διαχείριση. Επίσης είδαμε πώς προχωρούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς εντόπιζε συστήματα και εκπονούσε συστήματα. Πάντως βλέπουμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε και σε κάποια σύγκριση, όχι μόνο ιστορική αναδρομή από χρόνο σε χρόνο και τι αλλάζει. Μπορεί να αλλάζουν τα μέτρα και τα σταθμά, ο τρόπος που γίνονται οι μετρήσεις δεν θα πρέπει να είναι μόνο ποσοτικός. Άμα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ποιοτική βελτίωση, να μπορούμε και αυτή να τη μετρούμε. Στη συνέχεια, οι γενικές διευθύνσεις, ακούμε, σε αυτή την αναδρομή που κάνατε από το 2013 μέχρι το 2017 και τις συστάσεις που εφαρμόστηκαν. Τι βλέπουμε, ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές στη μεθοδολογία το οποίο μας δυσκολεύει επίσης να συγκρίνουμε τα πράγματα. Και όπως ε, και εσείς ο ίδιος είπατε, σας είναι δύσκολο ε, για το πώς μετρούν τα ασφάλματα ε, γενικές διευθύνσεις που έχει κάθε μία το δικό της σύστημα, κατάλαβα καλά. Λοιπόν, στην άμεση διαχείριση εκεί βελτιώθηκαν τα πράγματα και με ποιο τρόπο. Μιλήσατε και για την έμεση διαχείριση, δηλαδή με εξωτερική ανάθεση, με ε, ανάθεση που ε, στους αποκεντρωμένους οργανισμούς ή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όλα αυτά πώς τα εξετάζετε και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε μετά το 17, 18, 19 που έχει φτάσει ήδη. Αυτή την έμεση, επαναλαμβάνω, διαχείριση που υπερβαίνει το πλαίσιο, έτσι, το αμυγές των συστάσεων. για να υπάρχει και κάποια συνοχή εκεί και να μπορούμε να το παρακολουθούμε, να συγκρίνουμε και να μας χρησιμεύσει ως εργαλείο για να κάνουμε και καμία διόρθωση, με το μολύβι δηλαδή. Λέτε, και αυτό το μάθαμε και εμείς από το διάλογο αυτό που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ε, υπάρχει μια εστίαση ποσοτική. Στα διορθωτικά ταμεία που ήταν πολλά χρήματα, ε, ε, κάθε σφάλμα σήμαινε μεγάλο ποσό. Το ίδιο στην κοινή γεωργική πολιτική. Επειδή ήταν τεράστια τα ποσά, το παραμικρό σφάλμα ήταν μεγάλο ποσό. Τι γίνεται όμως με την ποιοτική ανάλυση, τα αποτελέσματα, ε, ιδιαίτερα από το 17 ας πούμε, ε, το θέμα της μετανάστευσης. Εκεί τι έχει γίνει. Η ποσότητα, το ποσό των χρημάτων δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά οι επιπτώσεις της καλής ή ε, κακής διαχείρισης μπορεί να είναι ολέθριες και καταστροφικές. Και απέναντι στους πολίτες. Πώς θα τα πούμε αυτά. Εσείς ως εσωτερικός ε, ελεγκτής, τα ξέρετε αυτά, τα έχετε δει από το 17 και μετά. Έτυχε να ακούσουμε εδώ, ε, στο Κοινοβούλιο, από τους Γενικούς Διευθυντές, ότι εγώ είμαι εντάξει πεντακάθαρο γιατί δεν τον βλέπω τον εσωτερικό ελεγκτή και δεν με έλεγξε το ελεγκτικό συνέδριο φέτο. Οπότε εντάξει, καθάρισα. Ε, δεν πάει έτσι. Είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι μόνο το ποσοτικό, το λογιστικό, είναι και το ποιοτικό και θα πρέπει όλα αυτά να προγραμματίζονται και να αξιολογούνται σωστά. Ο προπολογισμό δεν προστατεύεται μόνο από ανακτήσει χρημάτων, αλλά και με την προστασία των αποτελεσμάτων που το έχουμε υποσχεθεί εμείς και με σημαντικά έγγραφα ε, σε διοργανικές συμφωνίες. Και μετά οι γενικές διευθύνσεις δεν μπορούν αυτά να τα λεωποιήσουν. Ε, αυτά. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε. Ο κύριος Κράφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως ότι οι αλλαγές έχουν νόημα μόνο εφόσον σημαίνουν βελτιώσεις και όχι αλλαγή για την αλλαγή. Μιλήσατε για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκείνη τη συζήτηση είπατε ότι θα πρέπει η προσέγγιση να είναι πιο συνεπής και πιο εναρμονισμένη σε όλους τους τομείς πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλω να πω ότι κατά την άποψή μου, οι βασικοί δείκτες που μας επιτρέπουν να μετρούμε την πρόοδο σε διάφορους τομείς είναι ήδη εναρμονισμένοι σε κάποιο βαθμό. Εδώ αναφέρομαι ε, ε, ποσά ε, που είναι σε κίνδυνο στις πληρωμές και στο καθάριστο κλείσιμο των λογαριασμών. Έχουμε και αιτήσια πληροφόρηση για τα ποσά που κινδυνεύουν τη στιγμή που γίνεται η αιτήσια έκθεση πεπραγμένων. Συμφωνώ ότι περισσότερες γενικές διευθύνσεις δίνουν ε, επιπλέον δείκτες και πληροφόρηση για άλλες ιδιαιτερότητες των ε, δικών τους ε, τομέων αρμοδιοτήτων. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για να υπάρχει καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για την κατάσταση που επικρατεί στους διάφορους τομείς. Βεβαίως, πάντα χωράει βελτίωση και λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές σας ανησυχίες και άλλων μελήματα, έτσι ώστε να μπορούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι να κατανοούν τι συμβαίνει. Υπάρχουν όμως και όρια στο τι μπορεί κανείς να κάνει, διότι έχουμε διαφορετικό νομικό πλαίσιο, διαφορετικό οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο έχει ιδιαιτερότητες και πρέπει αυτές να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, τι συνέχεια θα δώσουμε σε τομείς που καλύπτονται από την ε, έμεση διαχείριση. Το, το ανέφερα και προηγουμένως. Οι αντιδράσεις, ε, και όσα ακούω από τις Κεντρικέ υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις επιχειρησιακές λειτουργικέ γενικές διευθύνσει Τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη και τώρα αναλύουμε ε, πώ θα συσταθεί μια μαθαργασία κεντρικέ κεντρικές υπηρεσίες, IS και ε, λειτουργικές επιχειρησιακές υπηρεσίες για να δούμε ε, από τις εκθέσεις ε, πώς θα εντοπίσουμε τις αδυναμίες για να ενισχύσουμε την ελεκτική διαδικασία και στο μέλλον αυτή η στενή παρακολούθηση των συστάσεων κατά τα άλλα συμβαίνει ήδη σε όλους τους άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τέτοια ε, υψηλά ποσοστά εκτέλεσης των προγραμμάτων δράσης που ακριβώς ε, καταρτίστηκαν για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που είχαμε εντοπίσει. Πρώτον, γενικά, περίπου το 100% όλων των συστάσεων είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν οι ελεγχόμενοι και τα υλοποιούν αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η παρακολούθηση αυτή είναι πάρα πολύ στενή, πάρα πολύ ε, λεπτομερής και ε, ε, υπάρχει και μια επιτροπή προόδου ε, του λογιστικού ελέγχου που μας βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όποτε έχουμε δυσκολίες, όπως έχουμε όποτε, κάποια συζητήσει με τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη αυτή Επιτροπή Ελέγχου της Προόδου ε, επεμβαίνει για να βοηθήσει να βελτιωθούν τα πράγματα με τον τρόπο που εμείς ε, τα προτείναμε. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας αν όχι, παρακαλώ να τις επαναλάβετε και ελάτε να σας ε, δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ έχω να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις. Ε, στην έκθεση αναφέρεται, γίνεται επανειλημμένα λόγος για αδυναμίες. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό, ποιες είναι αυτές οι αδυναμίες. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Μετά το δεύτερο αφορά την ίδια την έκθεση και τους ε, διεθνείς ε, χρηματοψηφιστικούς οργανισμούς, τους IFIS. Στην έκθεση λοιπόν ε, διαβάζω ότι η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ τις ε, προχρηματοδοτήσεις, ε, τις ε, διευκρινίζει και τις ελέγχει μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια τι μπορεί κανείς να ελέγξει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο η προστασία του προεπλογισμού, αλλά με ενδιαφέρει επιτόπου να υπάρχει κάποια πειθαρχία και κάποια αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 10 χρόνια τι μπορώ να κάνω. Και επ' αυτού τι έχετε να πείτε, τι, ισχύει τώρα κατόπιν με το Γενικό Γραμματικό, ε, και με τον κύριο Τιγκέρ μιλήσαμε για το Audit Progress Committee. Ε, ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και ρωτώ μια τέτοια επιτροπή. Τι είδους συμπεράσματα μπορεί να εξάγει από τα αποτελέσματα που παρουσιάζει κανείς σε αυτή την Επιτροπή. Και αναφέρεται ότι αυτή η Επιτροπή Πρόοδου του Ελέγχου ε, δεν είναι μια επιτροπή ε, σχετικά με την απόδοση της διαχείρισης, γιατί είναι και τελείως διαφορετικές πληροφορίες. Πληροφορίες που διοχετεύονται. Αλλά τώρα ακούμε ένα θόρυβο. Δεν ξέρω, ε, έχει κανείς ανοίξει την ηλεκτρική σκούπα, σκουπίζει. Ah ναι, Also, das, genau. Also, Leute, Leute, Leute. Ja, danke. Ähm, genau, also, <clears throat> also Audit Progress Committee war das eine, also Λοιπόν, ε, σας μίλησα για την Επιτροπή Ελέγχου του Πρόδου του Ελέγχου, ελέγχου της Πρόοδου. Ε, μετά υπάρχουν θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Υπάρχει ένα ερώτημα. Το Γιάσπερ και τα στοιχεία που δεν δίδονται από την ΑΙΠ κυρίως αναφορά αφορά τη σύγκρουση συμφερόντα. Δηλαδή η Γενική Διεύθυνση για τα περιφερειακά θέματα δεν παίρνει τα απαραίτητα στοιχεία, τότε νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί το πρόγραμμα. Μήπως μπορείτε να τοποθετηθείτε και από αυτού. Και κάτι άλλο. Η κυρία Επίτροπος, η κυρία Γεωργίευα ασχολείται με το θέμα των αποτελεσμάτων, budget for results. Ε, καλό που το θίξατε αυτό στην έκθεσή σας και θέλουμε να ξέρουμε τελικά ποιος παίζει ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτά που είπατε τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ρωτώ ε, κατά πόσον υπάρχει ε, ρόλος της Γενικής ε, με άλλα λόγια, πώς έχουμε προχωρήσει με αυτό το budget for results. Γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλετε να είμαι ήταν μόνο μία κίνηση ε, για επηρεασμό της κοινή γνώμης. Υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, χειροπιαστά. Και παρακαλώ έχετε το λόγο για να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε με τη σειρά που υποβάλλετε τις ερωτήσεις αυτές. Καταρχάς, με ρωτήσατε τι είναι οι αδυναμίες στις οποίες αναφερόμαστε στην έκθεση αυτή. Έχουμε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο τρόπο για να ταξινομούμε τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν από τους ελέγχους μας. Τα πορίσματα αυτά βαθμολογούνται τροποντινά και μπορώ να σε εξηγήσω πώς κατανομούμε τα πορίσματα αυτά. Μία σημαντική αδυναμία είναι θεμελιώδης αδυναμία η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις στο σύνολο ή σε ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας ελέγχου ή του υποκείμενου σε έλεγχο, για παράδειγμα μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική αδυναμία η οποία επηρεάζει το σύνολο μιας Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα στατιστικά δεδομένα τα οποία υποβάλλουμε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης θα έχετε δει ότι έχουμε έναν πολύ χαμηλό αριθμό συστάσεων που σχετίζονται με σημαντικά σφάλματα. Για μένα αυτό αποτελεί ένα σημαντικότατο δίκτυο ότι έχουμε τελικά ισχυρά συστήματα. Πάντω σαφώς αντιμετωπίζουμε τις σημαντικέ αυτές αδυναμίες όταν τις εντοπίζουμε. Παρέχουμε επίσης πληροφορίε όσον αφορά τις θεμελιώδεις αυτές αδυναμίες, αλλά και για τις πολύ σημαντικές τις λεγόμενες αδυναμίες, οι οποίες αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, αδυναμίες οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειε στο σύνολο ή σε μέρο τη διαδικασία ελέγχου. Δεν αφαιρόμαστε εδώ πέρα σε μια γενική διεύθυνση, αλλά σε μια διαδικασία ελέγχου. Και λέμε ότι μπορεί, μπορεί οι αδυναμίε αυτές να επηρεάσουν ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας ελέγχου και έπειτα περνάμε και σε περισσότερες λεπτομέρειε για το πώ θα πρέπει να περιγράφονται οι αδυναμίε αυτέ πότε θα πρέπει να εφαρμόσετε συγκεκριμένε συστάσει κ.ο.κ. Όσον αφορά τι σημαντικέ αυτέ κριτικέ, μάλλον θεμελιώδει αδυναμίε, τις πιο σημαντικές δηλαδή, για αυτές θέλουμε άμεση ανάληψη δράσης, προκειμένου τα κακό κείμενα να θεραπεύονται άμεσα. Όταν έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική σύσταση, προφανώς θέλουμε να έχουμε και μια άμεση αντίδραση. Και για τις σημαντικές αδυναμίες, και για αυτές θα πρέπει να έχουμε πάλι μια άμεση ανάληψη δράσης. Σας τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε λίγο πώς ταξινομούμε, πώς κατηγοριοποιούμε σε διαφορετικές κατηγορίες όλες αυτές τις λεγόμενες αδυναμίες. Όσον αφορά τώρα τα χρηματοπιστωτικά μέτρα και τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, συμφωνώ μαζί σα ότι όταν απαιτούνται 10 ολόκληρα χρόνια για να γίνει εκαθάριση μια διαδικασία προχρηματοδότηση, αυτό αποτελεί ασθενέ σημείο και το έχουμε εντοπίσει στην έκθεσή μα. Πρέπει όμω να λάβουμε υπόψη μα και ποιε είναι οι νομικέ απαιτήσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Ξέρω ότι μερικέ φορέ δεν είναι δυνατό να προβεί κανεί σε καθάριση μια προχρηματοδότηση νωρίτερα. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή Πρόεδρου του Ελέγχου, την APC. Σας είπα ότι η Επιτροπή αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει συμβουλές και ουσιαστικά εποπτεύει όλες τις δικασίες και όλα τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς κυρία Πρόεδρε αναφερθήκατε στα αποτελέσματα του ελέγχου μας όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου επικρίνεται εκεί ότι η έπιση δεν έλαβε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς οι υπεύθυνοι του διοικητικού ελέγχου αντιμετωπίζουν σημαντικές αδυναμίες και λέγεται επίσης ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι οριζόντιοι κίνδυνοι, οι εγκάρσιοι κίνδυνοι, αλλά ότι δεν προβλέπεται στην εντολή της Επιτροπής αυτής ότι θα πρέπει να ασχολείται με τους κινδύνους αυτούς. Και επίσης το Corporate Management Board δεν ασχολήθηκε με τους σημαντικούς κινδύνους σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων που δεν έχουν οριζόντιο ρόλο, μολονό ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στόχο διόρθωσης για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Corporate Management Board μέσω των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και των άλλων κεντρικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει παρόλα αυτά μια σφαιρική εικόνα όλων των σημαντικών κινδύνων, είτε αυτή είναι οριζόντι είτε μη οριζόντι. Στη συνέχεια το Corporate Management Board θα αποφασίσει για το αν απαιτείται να διεξαχθεί μια συζήτηση με τους αρμόδιους επικεφαλείς των γενικών διευθύνσεων και εν συνεχεία θα καταρτήσει ένα συγκεκριμένο κατάλογο όπου θα υπάρχουν και περαιτέρω πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μαζί με τον κατάλογο των σημαντικών κινδύνων φτάνουν σε εμά και στι υπόλοιπε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί στον δικό μα τον έλεγχο, λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία αυτά και ξέρετε ότι επί του παρόντο, κάνουμε μία στρατηγική ανάλυση κινδύνου για τα επόμενα τρία χρόνια. Θα λάβουμε λοιπόν υπόψη τι πληροφορίε αυτέ και φτάνουν πληροφορίες από διάφορες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες τροφοδοτούνται στη συνέχεια στην ε, APC. Η Audit Progress Committee λοιπόν λαμβάνει πληροφορίες από το ε, Corporate Management Board για όλους τους κινδύνους αυτούς οι οποίοι θεωρούνται οριζόντιοι και μη και εν συνεχεία η APC μπορεί να δει αν υφίστανται κενά ανάμεσα στην αξιολόγηση του κινδύνου και την δράση που ανέλαβαν οι υπεύθυνοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιολογεί επίσης τον κίνδυνο και αξιολογεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει τους κινδύνους αυτούς. Και αφού κάνει τις αξιολογήσεις αυτές, η APC μπορεί να προβεί σε περαιτέρω δράση στην πράξη μπορεί να μας πει ότι πρέπει να αναλάβουμε περαιτέρω δράσεις ή μπορεί να έρθει σε επαφή ακόμα και με το Corporate Management Board για να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Όσον αφορά το Γιάσπερ, όντως εντοπίσαμε προβλήματα με το πρόγραμμα αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να μην πω αδύνατο να καταφέρουμε να αναλύσουμε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα Τη ε, εφαρμογή των διαφόρων δράσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του Γιάσπερ. Στο σχέδιο δράση πάντω το οποίο υποβάλαμε, προβλέπουμε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τον προπολογισμό, ο οποίο θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων, budget for results, θα ήμουν πιο αισιόδοξο από εσά, κυρία Πρόεδρε, διότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση διάβασα στην ετήσια έκθεση επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο ίδιος ο ΩΣΑ θεωρεί ότι το πλαίσιο επιδόσεων μας είναι ισχυρότερο από το πλαίσιο επιδόσεων οποιοδήποτε κράτους μέλους του ΩΣΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι, αλλά σίγουρα καταδεικνύει ότι ήδη έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα και αν ανατρέξετε τις διάφορες εκθέσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει και τις οποίες έχουν υποβάλει και μεμονωμένες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να λάβετε πάρα πολλές θετικές πληροφορίες για τα θετικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε επιτύχει. Προφανώς προκύπτουν κάποια ζητήματα και δυναμίες. Την τελευταία φορά θυμάστε ότι συζητήσαμε το ζήτημα των στατιστικών δεδομένων εκείνων που δεν υποβάλλονται που δεν καταρτίζονται μάλλον από τη Eurostat. Στην περίπτωση αυτή όντω υπήρχαν κάποιες αδυναμίες ακριβώς επειδή ο έλεγχος της ποιότητα δεν είναι στο επίπεδο εκείνο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει η Eurostat. Εγώ λοιπόν θα ήμουν πιο θετικός και αισιόδοξο όσον αφορά το budget for results και ιδίω αν δείτε για τα σχέδια δράσης ε, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις ε, όσον αφορά τους ε, επιμέρους τομείς στους οποίους κάνουμε ελέγχους επιδόσεων, τότε βλέπετε εκεί ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης κατάστασης στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα. Μάλιστα. Τώρα να μην τα ανακατέψουμε αυτά τα δύο ε, για την Επιτροπή Προόδου που πολύ ωραία το εξηγήσατε, ε, για εκείνο που σας ανέφερα προηγουμένως, για την ιεράρχηση των προβλημάτων. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω όμως εγώ. Σε αυτή την ιεράρχηση, όπου κοιτάτε αν ένα πρόβλημα και το εντοπίζετε, αν αφορά όλο το θεσμικό όργανο ή απλώς μια διαδικασία ή ένα σύνολο διαδικασιών, με ποιο τρόπο βρίσκεται ποιος είναι αρμόδιος και υπεύθυνο το πρόσωπο που χρειάζεται να λύσει το πρόβλημα. Και μιλήσατε και για ένα χρονοδιάγραμμα. Πώς ορίζεται αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ποιος το ορίζει, εσείς ο ίδιος. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή ποιος το χαρακτηρίζει αν είναι επίγον ή λιγότερο επίγον. Λοιπόν, πρώτον, πώς βλέπετε, πώς καταλαβαίνετε ποιο είναι ο υπεύθυνο και πώς ε, χαράζεται ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυσή του. Για να καταλάβουμε λίγο πώς ε, λειτουργούν αυτά τα πράγματα και στην άμεση και στην έμεση διαχείριση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κύριο κύριος Κράφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στους εσωτερικούς ελέγχους που κάνουμε, τις λογιστικούς και τις εκθέσεις μας, σαφώς αναφέρουμε τη φύση του ευρήματος. Αν είναι κρίσιμο, πολύ σημαντικό, σημαντικό. Καθώς επίσης και ε, τη σύσταση που συνδέεται με αυτό και την προτείνουμε εμείς για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό το συζητούμε με τον ελεγχόμενο και θα πρέπει ο ελεγχόμενος να εξηγήσει ακριβώς ποια δράση σκοπεύει να ε, λάβει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εμείς εντοπίσαμε και ο ίδιος θα μας πει και μια προθεσμία, μια καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι πότε θα το έχει κάνει. Εάν δεν μας ικανοποιεί η απάντηση, είτε το χρονοδιάγραμμα, είτε η λύση που προτείνει, η δράση δηλαδή που προτείνει, αν θεωρήσουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα, δεν θα δεχτούμε το πρόγραμμα δράσης. Αν θεωρήσουμε επίσης ότι κάτι τραβάει πολύ σε μάκρος για να εφαρμοστεί ή για να διορθωθεί, πάλι θα πούμε ξεκάθαρα ότι δεν δεχόμαστε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Σας είπα ότι για το 99% όλων των συστάσεων που κάνουμε, ε, γενικά συμφωνούμε με το προτινόμενο πρόγραμμα δράσης. Πρέπει όμως να ε, ομολογήσω επίσης ότι όποτε υπάρχει θέμα, όχι πολύ συχνά, όταν ένας ελεγχόμενος δεν δέχεται μια σύσταση, υπάρχει η τάση, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πρόοδο του Ελέγχου ε, υπάρχει περίπτωση να τον καλέσει να έρθει στην Επιτροπή και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν δέχεται τη σύσταση. Αυτό το έχουμε δει σε δύο περιπτώσεις ε, που δεν ε, συμφωνούσε ο ελεγχόμενος με τις δικές μας συστάσεις. Ε, γιατί ας πούμε δεν είχε τους απαραίτητους πόρους, είχε κάποιους άλλους περιορισμούς και διαφώνησε με τη δική μας σύσταση. Σε δύο περιπτώσεις λοιπόν δεν έχουμε συμφωνήσει. Σε όλες τις υπόλοιπες, σας είπα το 99% ε, συμφωνούν απολύτως. Και μετά υπάρχει και η ε, εκτέλεση, η υλοποίηση των δράσεων, όπου παρακολουθούμε εμείς πολύ στενά τι γίνεται. Έχουμε μια βάση δεδομένων ε, όπου δηλώνει ο ελεγχόμενος τι δράσεις υλοποιεί σε ποιο χρονικό πλαίσιο και βάσει αυτών κάνουμε και ε, την παρακολούθηση. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι το κλείνουμε αυτό, το κλείνει τη σύσταση. Θεωρούμε ότι έχει οθετηθεί. Αλλιώ επανερχόμαστε μέχρι να ε, γίνει σωστή διαχείριση. Θυμίζω ότι έχουμε 12 συστάσεις από όλο το μεγάλο αριθμό που σας ανέφερα όπου υπήρξε καθυστέρηση άνω του εξαμήνου ακόμα και σε αυτή την περίπτωση συνεχίζουμε ε, για να βεβαιωθούμε ότι αναλαμβάνεται δράση. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα ότι οι μισές από τις 12 αυτές δράσεις που καθυστέρησαν για μεγάλο διάστημα τώρα εφαρμόζονται. Και θα πιώσουμε, πιέσουμε μαζί με την ε, Επιτροπή Ελέγχου, του πρόοδου μάλλον του ελέγχου, να το υλοποιήσουν και οι υπόλοιπε γενικές διευθύνσεις. Ακριβώς. Έχω και εγώ ερωτήσεις που ε, ταιριάζουν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Έχω εδώ τις συστάσεις για το Τζάσπερ και τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Πολιτικής. Τι έχει αλλάξει εκεί ε, στην πρόσβαση του ε, EAS. Για να καταλάβω, άλλαξε τίποτα στο Τζάσπερ όταν κάνετε συστάσεις. Και μετά τι έχει αλλάξει στην τακτική της ΤΕΦΚΟ για τις προκαταβολές. και το τρίτο που το είχα ξεχάσει μέχρι τώρα, τα στατιστικά στοιχεία. Επικρίνεται το θέμα των, ε, της αξιοπιστίας των στατιστικών που έχουν γίνει εκτός Eurostat. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Γενική Διεύθυνση Grow και εκείνους που πρέπει να παρακολουθούν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η κριτική σας σε τι αναφέρεται ακριβώς και τι έχει αλλάξει εκεί ή τι πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το Jaspers ε, το σύστημα, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες ε, ε, στο, στη σελίδα 58 της Staff Document της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. συστήνουμε στην Γενική Διεύθυνση Περιφέρειες να εξετάσει λίγο τις δραστηριότητες του Jaspers, να κάνουν επιτόπου ελέγχους όσον αφορά τις, τους εσωτερικού ελέγχους του Jaspers και επίσης να ελέγξουν και το εσωτερικό σύστημα ελέγχου του JASPERS. Επίσης προτείνουμε μία μέσο μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του συστήματος όπως αναφέρεται στο 2.4 ε, της συμφωνίας, ε, πλαίσιο, συμφωνίας πλαίσιο συνεργασίας έτσι ώστε να ε, εντοπιστούν κάποια συγκεκριμένα εργαλεία και η Γενική Διεθνή Ρίτζο θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει και τα δικαιώματα πρόσβασης που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα Jaspers, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης σε συστήματα ενημέρωσης, σε έγγραφα, σε αρχεία που έχουν σχέση με τους ελέγχους. Ε, τελική έκθεση και με βάση το πρόγραμμα δράσης που συμφωνήθηκε ε, έλαβαν, υλοποιήθηκαν από τη Ρίτζο συγκεκριμένες δράσεις σε στενή συνεργασία με το σύστημα Jaspers έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση σημαντικών προγραμμάτων κυρίως για να υπάρξει καλύτερος ορισμός των ε, συμβασιακών υποχρεώσεων και να υπάρχει και εποπτεία του συστήματος αξιολόγησης του Jaspers και επίσης και για να περιστεί οποιοδήποτε κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει ανάμεσα ε, στο σύστημα, στα συστήματα που εφαρμόζει το Jaspers. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι τώρα δεν έχουμε ε, παρακολουθήσει την εξέλιξη όλου αυτού, αλλά θα επανέλθουμε για να σας ενημερώσουμε για το ποιες είναι οι θετικές ε, τα θετικά συμπεράσματα που ενδεχομένως έχουν προκύψει από τις δράσεις που έχουν μεταξύ αναπτυχθεί. Όσον αφορά τώρα την ΤΕΦΚΟ. Ίσως τώρα αυτά που θα πω να είναι τεχνική φύσεω. Γνωρίζετε το clearing μπορεί να γίνει μόνο με πάνω στη βάση των πληροφοριών για τις πραγματοποιητήσεις δαπάνες. Άρα πρέπει να υπάρχουν πραγματικές δράσεις που να αναπτύσσονται επί τόπου και να προκύπτουν σχετικές δαπάνες. Αυτά υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δημοσιονομικά εργαλεία δεν έχουν όλα τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτές τις πληροφορίες πριν κλείσει, πριν ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. Και μερικές φορές έχετε δίκιο, τα προγράμματα είναι μακροχρόνια. Τώρα έχουμε το νέο δημοσιονομικό οργανισμό που προβλέπει μια καινοτομία. Λαμβάνεται αυτό υπόψη και η τελική εκαθάριση γίνεται το αργότερο όταν ολοκληρώνεται, λίγο πριν μάλλον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αυτό είναι μια νέα νομική προϋπόθεση που είναι ενσωματωμένη στο νέο χρηματοδοτικό κανονισμό και θέλουμε αυτό να εφαρμόζεται από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ μαζί με την IFIs. Δεν απαντήσετε για το θέμα των ε, στατιστικών δεδομένων. Ε, πράγματι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω το εξής κάναμε έναν έλεγχο για τα στατιστικά δεδομένα που υποβάλλει η ίδια η Eurostat. Και με λίγα λόγια, το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι η έκθεση ελέγχου πρόοδου είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Άρα το σύστημα είναι ικανοποιητικό. Τα στατιστικά δεδομένα της Eurostat από με αυτά των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών είναι αξιόπιστα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια τα δεδομένα σε διάφορους άμεσα ενδιαφερόμενους. Όσον αφορά όμως στατιστικά δεδομένα που δεν είναι της Eurostat, εκεί διαπιστώθηκε ότι το σύστημα δεν είναι αρκετά στεγανό. Η η Γενική Διεύθυνση ε, Eurostat δέχτηκε τις συστάσεις και τώρα συνεργάζεται με όλες τις κεντρικές υπηρεσίες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και θέλω να αναφερθώ στη δέσμη μέτρων διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως γνωρίζετε εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2018. Εκεί προβλέπεται η ενίσχυση του Corporate Management Board αλλά και η διαχείριση των δεδομένων και αυτή λαμβάνεται υπόψη σε, αυτό, σε αυτή τη δέσμη μέτρων διαχείρισης. Υπάρχει μια υπομάδα ε, της ε, εταιρικής ομάδας διαχείρισης του Corporate Management Board ε, που εξαρτώνται από τα στατιστικά δεδομένα που δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί λοιπόν έλαβαν υπόψη τους το πρόγραμμα δράσης το οποίο δεχτήκαμε εμείς δέχτηκαν τα δεδομένα για να μπορούν να προβούν σε ενέργειες και να μειώσουν κινδύνους σε σχέση με δεδομένα, στατιστικά πάντα δεδομένα που δεν υποβάλλονται από τη Eurostat. Πρόεδρος, ξέρω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά προηγουμένως ε, ε, θίξατε τη συζήτηση για το νέο πρόγραμμα στον γεωργικό τομέα. Υπάρχει λοιπόν το εξής ερώτημα όσον αφορά τους δικαιούχους. Ε, ξέρουμε ότι εσείς δεν έρχεστε σε επαφή με τους δικαιούχους. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Έχετε κάνει κάποιες συστάσεις για αυτά τα προγράμματα για να γνωρίζουμε τι γίνεται τελικά με τους τελικούς δικιούχους ε, τόσο στα, από τα διαρθρωτικά ταμεία όσο και από γεωργικές παροχές. Όχι, δεν έχουμε καταθέσει καμία πρόταση που να αφορά στις ε, νομικές ε, προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί σε εσά και στο Συμβούλιο. Αλλά Βεβαίως, οι εκθέσεις μας ελέγχου περιλαμβάνουν συστάσεις που εξετάζουν κάποιες αδυναμίες των ε, συστημάτων που είχαμε εντοπίσει παλαιότερα. Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσον μεταβαίνουμε επιτόπου και κατά πόσον ερχόμαστε σε επαφή με τον τελικό δικαιούχο, είναι αλήθεια ότι αυτό εμείς δεν το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να είναι συγκρίσιμος με αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά καιρού όμως, ε, αν αξιολογούμε τη δουλειά που κάνουν οι Γενικές Διευθύνσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ο δικός μας λοιπόν ο στόχος είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσον ε, λειτουργούν σωστά οι γενικές διευθύνσεις, ε, ε, κατά πόσον λειτουργούν τα συστήματα στα κράτη-μέλη, μέχρι και στον τελευταίο δικαιούχο. Και εμείς φέρουμε την ευθύνη, ε, οι συνάδελφοί μας συγκεκριμένα, να μεταβούν επιτόπου για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς λειτουργούν οι εθνικές αρχές εμείς τους ε, συνοδεύουμε για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα της ε, δουλειάς. Αυτά λοιπόν όλα τα κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που να μας προσφέρει ε, τη σιγουριά ότι τα συστήματά μας ελέγχου είναι αποτελεσματικά ή όχι. Εμείς όμως ε, όπως σας είπα, ε, δεν ερχόμαστε σε τελική επαφή, σε επαφή με τον τελικό αποδέκτη, τον τελικό δικαιούχο. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε, να πηγαίνουμε επί τόπου, αλλά σας είπα, εμείς ε, επί τόπου κάνουμε αυτά που σας παρουσίασε μόλις πριν από λίγο. Τα περισμένα χρόνια ο εσωτερικός ελεγκτής εργάστηκε πάρα πολύ σε θέματα διαφάνειας στο γεωργικό τομέα κυρίως και λιγότερο στα διορθωτικά ταμεία για τα διορθωτικά μέτρα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ε, σε ό,τι αφορά τις κοινοποιήσεις των οργανισμών πληρωμών. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν σαφείς οι συστάσεις και πολύ μεγάλες διορθώσεις που έγιναν. Τώρα πώς έχει η κατάσταση, είναι πιο διαφανής, πιο αξιόπιστη, είναι αρκετά αυτά που κάνουν γενικές διευθύνσεις και στη Γεωργία και στην περιφερειακή πολιτική. Με βάση ε, τις εκθέσεις ε, οικονομικού ελέγχου που κάναμε για τη συνδιαχείριση ε, της, της συνοχή και στη Γεωργία, λειτουργεί το σύστημα βεβαίως, αλλά δεν είναι ένα σύστημα μηχανικό στατιστικό. Δηλαδή, εάν τα κράτη-μέλη εργάζονται σωστά, τότε έχουμε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα. Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους τα κράτη-μέλη, τότε εμεί κάνουμε προσαρμογές, αλλά αυτό δεν γίνεται με μια στατιστική βάση. Αυτό πρέπει να βασίζεται στην επαγγελματική αξιολόγηση και κρίση. Οι συνάδελφοι λοιπόν στις διάφορες επιχειρησιακές γενικές διευθύνσεις αναλύουν τις αδυναμίες που υπάρχουν έτσι ώστε να εκτιμούν ποιο θα είναι ε, το ο αξιόπιστο ποσό σε κίνδυνο που παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα το βρείτε ως πληροφορία στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων ε, των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Όπως σας είπα, η γενική γνώμη που έχω δώσει εγώ ε, για την οικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή βασίζεται σε αυτό. Και το εξή είναι απολύτως βέβαιο. Ο προπολογισμό προστατεύεται συνολικά και με την πάροδο του χρόνου. Εάν συγκρίνεται το κίνδυνο στις πληρωμές και τις διορθώσεις που καλούνται να εφαρμόσουν τα διάφορα κράτη στους διάφορους τομείς, τότε είναι σαφές ότι ε, είμαστε πολύ πιο κάτω από το όριο του στατιστικού λάθους του 2%. Βεβαίω έχουμε τη γνωμοδότηση, ε, ταυτόχρονα υπάρχουν δυνατότητες και ανάγκες, καμιά φορά βελτιώσεων, που εγγράφονται στις επιφυλάξεις που βάζω και στη γενική μου γνωμοδότηση. Λειτουργεί το σύστημα, αλλά όπως σας είπα, δεν είναι τέλειο. Πάντα χωράει βελτίωση. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι και στο μέλλον θα είναι θετική η επίπτωση και ο αντίκτυπος. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, έλεγα ότι ήθελα να ρωτήσω τον κύριο. Στον οποίο αναθέσατε να ασχοληθεί αυτά τα θέμα, με τα θέματα λόγω σύγκρουση συμφερόντων δικό σα. Ε, ξέχασα και το όνομά του και ζητώ. Είναι ο κύριο Τζεφ Μέισον. Ζητώ συγγνώμη κύριε Μέισον, μου διέφυγε το όνομά σα. Όπω Όπως εξηγήσε και ο Μάντφρετ, Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα προκειμένου να αποφύγουμε τις αδυναμίες αυτές στην πράξη. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι το τελευταίο, το τελευταίο έτος και κάποιους μήνες έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους για τις ανακτήσεις κονδυλίων, καθώς επίσης και την οικονομική αποδοτικότητα των ελέγχων και επίσης ο μεγάλος έλεγχος στον οποίο αναφέρθηκε ο Μάνφρετ όσον αφορά το σύστημα αυτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα απασχόλησε πάρα πολύ τελευταίο έτο και οδήγησε σημαντικέ αλλαγέ. Στην περίπτωση αυτή, ο Μάνφρετ και εγώ συνυπογράφουμε τελική έκθεση. Αυτή είναι η βασική κέρυη τομή επί τους οποίους, για τους οποίους υπήρξε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Μάνφρετ ασχολήθηκε με ένα τμήμα του ελέγχου και συνυπογράψαμε έπειτα την τελική έκθεση που αναφέρεται στο σύνολο των ελέγχων αυτών που διεξήχθησαν. Ωραία, δεν ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Ολοκληρώθηκε εδώ το συγκεκριμένο σημείο τη μέρη τη διάταξη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ άξιζε πάρα πολύ το κόπο που βάλαμε ξανά το θέμα στη μέση διάταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλο το έργο αυτό που κάνετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας σε αυτό το τομέα που για μας είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σημείο ε, 8 της ημερησίας διάταξης. Ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ΑΙΟΠΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Η κυρία Κάντεμπαχ είναι ε, η συγγήτρια και από το ε, ελεγκτικό συνέδριο ο κύριος Σάτζιου, στον οποίο και δίνω μέσα το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χάρη στην ε, τεχνολογία μπορώ να προβάλλω και την παρουσίασή μου αυτή. Θα ήθελα καταρχάς να σε ευχηθώ όμως ένα ευτυχισμένο και ιδίως ιδιαίτερα επιτυχές 2019 και ιδίω αναφέρομαι σε αυτού οι οποίοι πρόκειται να επανεκλεγούν μετά τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, Σα εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Μπορούμε να δούμε τώρα τι διαφάνειε, παρακαλώ. Ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο για την ειδική αυτή έκθεση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να δούμε πώς λειτουργεί μία από τις βασικές αυτές υπηρεσίες, ένας βασικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να δούμε περισσότερο πώς λειτουργεί εν γέννη ο ασφαλιστικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θελήσαμε να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσατε εσείς ε, να, να ε, χρησιμοποιήσετε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των ε, ελεγκτικών εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε στη διαφάνεια αυτή ότι ε, κατά μέσο όρο το ποσοστό των ασφαλίστρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το ΑΕΠ δεν είναι τόσο εντυπωσιακά σε σχέση με άλλους τομείς. Είναι περίπου ένα 19% του ετησίου ΑΕΠ των ε, μεμονωμένων κρατών μελών. Υπάρχει όμω εδώ πέρα μεγάλη απόκληση και πολλές διαφορές. Τα αποτελέσματα είναι άνισα αυτή τη στιγμή και προκύπτουν και διάφορα διασυνοριακά ζητήματα, ένα ακόμα ζήτημα το οποίο μα απασχόλησε κατά τη διάρκεια τη έκθεση αυτής. Βέβαια, τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ασφαλίζει ο ασφαλιστικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, μιλάμε για πολύ σημαντικά χρηματικά ποσά. Τώρα, ποιο ήταν το πεδίο εφαρμογή αυτή τη ειδική έκθεση. Θέλαμε καταρχά να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όντω συμβάλλει στην λεγόμενη εποπτική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα συνεργαστήκαμε επίσης και με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Δεν είχαμε άμεση συμμετοχή των ε, εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Πάντω, τα πορίσματα θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να πούμε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί το πιο σημαντικό ζήτημα ή η πιο σημαντική ανησυχία, αν θέλετε. Υπάρχουν όμως δύο πτυχές στο ζήτημα αυτό, τις οποίες ε, ελέγξαμε. Καταρχάς, η ομοιόμορφη προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του ασφαλιστικού τομέα, που τελικά αφορά σχεδόν τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη, να έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση των καταναλωτών. Από την άλλη, ασχοληθήκαμε και με το ζήτημα του θεμητού ανταγωνισμού. Υπάρχει άραγε θεμητό ανταγωνισμό ανάμεσα στι διάφορε ασφαλιστικέ επιχειρήσει και πώ διασφαλίζεται αυτό. Εξετάσαμε λοιπόν πολλέ διαφορετικέ πτυχέ. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά συμπεράσματα. Α περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ποιο είναι το, ποια είναι τα γενικότερα συμπεράσματά μα. Η ΕΙΟΠΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλή και Επαγγελματικών Συντάξεων, συμβάλλει σαφώ στην εποπτεία και τη σταθερότητα του ασφαλιστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδρύθηκε το 2011, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, μετά την σημαντικότερη χρηματοπιστωτική κρίση που γνωρίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή δηλαδή του 2008-2009. Η ΕΙΟΠΑ λοιπόν είναι ένας, μία από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές που προέκυψε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση Πρόκειται για μια αρχή που πολύ ορθά αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτε ότι θα πρέπει να συσταθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενε μελλοντικέ οικονομικέ κρίσει. Μολονότι λοιπόν ο αρχικό τη ρόλο είναι πολύ σημαντικό, παρόλα υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία τη ΕΙΟΠΑ. Όχι επειδή η ΕΙΟΠΑ ω οργανισμό δεν είναι καλή ποιότητα, όχι επειδή υπάρχουν θέματα κακοδιαχείρισης, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα συστημική φύση κάτι το οποίο εμποδίζει την ορθή λειτουργία του εποπτικού αυτού οργανισμού είναι ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη διακυβέρνηση, δεν υφίστανται οι κατάλληλοι ανθρώπινοι και χρηματικοί πόροι και επίσης θα έλεγα ότι ε, το πιο σημαντικό τεχνικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη και απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών και τη ΕΙΟΠΑ. Ξέρετε ότι οι εθνικέ αρμόδιε αρχέ είναι παρούσε σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικέ αρμόδιε αρχέ συνεργάζονται με την ΕΙΟΠΑ για τη διασφάλιση τη σταθερότητα και τη εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα. Δεν έχουμε ενιαίο ασφαλιστικό τομέα ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέχουμε από ακόμη πολύ από την επίτευξη του στόχου αυτού. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίω με εμά, δηλαδή με του αρμοδίου στα κράτη-μέλη. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίω στι εθνικέ αρμόδιε αρχέ και δυστυχώς οι εθνικές αυτές αρμόδιες αρχές δεν συμβάλλουν αρκετά ώστε να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός εποπτικός έλεγχος όσον αφορά τον ασφαλιστικό τομέα. Θεωρώ λοιπόν ότι ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές μπορούν να υπερκεραστούν και ήδη έχουν ε, αντιμετωπιστεί εν μέρη από την ΕΙΟΠΑ, εμείς προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς εθνικές αρμόδιες αρχές, αλλά και προς εσάς, τους ε, νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είστε η μία σημαντική νομοθετική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθυνόμενοι λοιπόν και σε εσά, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Τώρα, τα εποπτικά εργαλεία. Τα εποπτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΟΠΑ. Αυτό είναι ένα τομέα που ελέγξαμε λίγο περαιτέρω. Εν θεωρούμε ότι τα εποπτικά αυτά εργαλεία λειτουργούν σωστά. Παρ' όλα αυτά, τα εποπτικά αυτά εργαλεία δεν είναι αρκετά στοχευμένα. Η σχετική μας λοιπόν σύσταση είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση των εποπτικών εργαλείων προκειμένου να μην έχουμε πορίσματα ιδιαίτερα γενικόλογα και προκειμένου τελικά να ενταθεί και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρμόδιες αρχές. Θέλουμε εδώ μεγαλύτερη στόχευση. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ελέγξαμε ήταν η διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, ζήτημα το οποίο θα ήθελα να τονίσω λίγο περισσότερο στην παρουσίασή μου αυτή. Όπως βλέπετε και σε αυτή τη διαφάνεια αλλά και στι προηγούμενες διαφάνειες υπάρχει μια άνηση θα λέγαμε κατανομή των ασφαλίστρων από την μία χώρα στην άλλη, πράγμα το οποίο έχει να κάνει καταρχάς με τον διασυνοριακό, τη διασυνοριακή φύση του επιχειρηματικού αυτού κλάδου. Και θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα και αν θέλετε με έναν τρόπο ιδιαίτερα χειρό ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της ενιαίας εσωτερική αγοράς είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της εσωτερική αγοράς. Στον πολύ ευαίσθητο όμως αυτό το τομέα, τον τομέα των ασφαλίσεων δηλαδή, εντοπίσαμε κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορούν απλώς να αντιμετωπιστούν από τους μεμονωμένους υπεύθυνους φορείς. Και αυτό διότι η υφιστάμενη αρχιτεκτονική παροχής διασυνοριακών ασφαλιστικών υπηρεσιών ουσιαστικά κατανέμει άνισα το βάρος ανάμεσα στις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές. Θα έλεγα ότι το πεδίο εφαρμογή εδώ πέρα είναι ιδιαίτερα ευρύ. Έχουμε πολύ σημαντικά ασφάλιστρα 110 δισεκατομμύρια σε ορισμένες χώρες που αντιστοιχούν στο 8% των συνολικών ασφαλίστρων που καταβάλλονται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Σε άλλες χώρες πάλι τα ασφάλιστρα είναι πολύ πιο χαμηλά. Μέσω της επόμενης διαφάνειας μπορούμε να δούμε πως την χάνει εποπτείας και ελέγχου η διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αν έχουμε μία μητρική ασφαλιστική εταιρεία που έχει θηγατρικές σε ορισμένες άλλες χώρες, τότε προβλέπετε εδώ ότι μπορούμε να έχουμε αυτό το οποίο στα αγγλικά ονομάζεται College of Supervisors, ένα συλλογικό εποπτικό όργανο στο οποίο συμμετέχει και η ΟΠΑ. Τα συλλογικά αυτά όργανα εποπτείας απαρτίζονται από την ΕΙΟΠΑ και από όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Κράτη-μέλη στα οποία έχει επιχειρηματική δραστηριότητα μια ασφαλιστική επιχείρηση. βασικός ρόλος των συλλογικών αυτών εποπτικών φορέων είναι να παρακολουθούν, να εποπτεύουν και να ελέγχουν τη διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αν δούμε όμως τους γενικότερους κανόνες που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, συντοποιούμε ότι ε, οι εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η μητρική επιχείρηση είναι αυτές οι οποίες έχουν τον πρωταρχικό ρόλο και βλέπουμε ότι τελικά επιβάλλεται εδώ περισσότερο η εθνική νομοθεσία και οι εθνικές αρμόδιες αρχές ή μάλλον η εθνική αρμόδια αρχή σε αυτό το κράτος μέλος ενδιαφέρεται περισσότερο για την οικονομική σταθερότητα της συγκεκριμένης χώρας αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ασφαλιστική αυτή επιχείρηση. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορε εθνικέ αρμόδιε αρχέ, καθώ επίση και με την ίδια την ΕΙΟΠΑ, ιδίω για το ζήτημα τη διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, και είδαμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει παρέχονταν πολύ χαμηλά ασφάλιστρα και αυτό αποτελούσε κίνητρο προκειμένου να πτυχθούν συγκεκριμένε επιχειρήσεις πάρα πολύ γρήγορα και κατά τρόπο αθέμητο τελικά σε ορισμένες χώρες. Δυστυχώ αυτό δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για την εποπτεία συγκεκριμένων εθνικών αρμόδιων αρχών. Μετά την παρέμβαση της ΕΙΟΠΑ, η οποία εκτελεί έναν έλεγχο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συνειδητοποίησαμε ότι υπήρχαν ορισμένε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αποκρύψει το γεγονός ότι βρισκόντουσαν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και πολλές φορές στο χείλο της χρεοκοπία. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι τονίζεται ακόμα περισσότερο η σημασία του ρόλου τη ΕΙΟΠΑ, η οποία θα, πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει και σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να εντοπίζει κατά αυτόν τον τρόπο τα κακό κείμενα. Στην επόμενη διαφάνεια εστιαζόμαστε σε έναν άλλον τομέα όπου βρίθουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Έχουμε τα λεγόμενα εσωτερικά μοντέλα. Πρόκειται για μοντέλα τα οποία ακολουθούν πολύ σημαντικές μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν πολύ πολύπλοκα ασφαλιστικά προϊόντα και οι οποίες ακολουθούν τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες ελέγχου και αξιολόγησης του κινδύνου ουσιαστικά θεσπίζουν ένα δικό του εσωτερικό σύστημα ελέγχου για να ελέγξουν τη δική τους οικονομική κατάσταση. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι δίκαιο και θεμητό. Στο ερώτημα αυτό μπορούν να απαντήσουν μόνο οι εθνικές αρμόδιες αρχές, οι οποίες καλούνται σε ένα πρώτο επίπεδο να ελέγξουν αυτά τα εσωτερικά μοντέλα ελέγχου. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμω είναι ότι τα εσωτερικά μοντέλα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφορά και μεγάλες αποκλίσεις από, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και βλέπουμε ότι ακολουθούνται αυτή τη στιγμή 200 διαφορετικά ιστορικά μοντέλα για τις χίλιες περίπου ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ η ΕΙΟΠΑ καλείται να συνδράμει τις εθνικές αρμόδιες αρχές προκειμένου με έναν ομοιόμορφο τρόπο να εποπτεύουν τα ιστορικά αυτά μοντέλα προκειμένου η ελοχεύονται κίνδυνοι να μπορούν να αξιολογούνται ομοιόμορφα και αντικειμενικά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στο πλαίσιο ενός μεμονωμένου κράτους μέλους. Η ΕΙΟΠΑ προσπάθησε να συνδράμει κατά αυτόν τον τρόπο τις εθνικές αρμόδιες αρχές αλλά αντιμετώπισε και αυτόν ιδιαίτερα ενδιαφέρον διάφορα εμπόδια. Και ουσιαστικά το πιο σημαντικό εμπόδιο ήταν ότι οι εθνικέ αρμόδιε αρχέ δεν επιθυμούσαν να ανταλλάξουν πληροφορίε με την ΕΙΟΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχει η ΕΙΟΠΑ μεγαλύτερη πρόσβαση στι πληροφορίε των εθνικών αρμόδιων αρχών. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε να το επιλύσετε το πρόβλημα αυτό. Ο υφιστάμενος κανονισμός προβλέπει ότι η ΟΠΑ έχει λίγα μόνο δικαιώματα προκειμένου πολύ ευγενικά να αιτηθεί από τις εθνικές αρμόδιες αρχές να τις παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικούς φορείς του ασφαλιστικού τομέα προκειμένου να του ζητήσει πληροφορίες. Με άλλα λόγια η ΕΙΟΠΑ δεν δύναται, δεν μπορεί και δεν προβλέπεται αυτό από την κοινωνική νομοθεσία να έρθει σε επαφή με συγκεκριμένες ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις προκειμένου να του ζητήσει πληροφορίες. Καταλαβαίνετε ότι αν η ΕΙΟΠΑ δεν έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία χρειάζεται, το σύστημα εποπτείας το οποίο πρεσβεύει ο οργανισμό, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ευοδοθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν εσεί οι νομοθέτε να τροποποιήσετε την αλόγω τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Πολύ γρήγορα. Όσον αφορά τι δοκιμέ αντοχή του ασφαλιστικού τομέα. Είδαμε ότι η δοκιμή αυτή αντοχή που χώρα το 2016 έδωσε θετικά αποτελέσματα. Εντοπίσαμε βέβαια και κάποιε αδυναμίε, αλλά το πιο σημαντικό πόρισμα θα έλεγα είναι ότι ε, επί του παρόντος, και αναφέρομαι εδώ πέρα στη δοκιμή εντοχής που έγινε το 2016, βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε μία γενική εικόνα της κατάστασης. Αυτό το οποίο ζητάμε και αυτό αποτελεί μέρο και των συστάσεών μα, και βέβαια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά μπορεί να γίνει κατεθελούσιο τρόπο. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι μεγάλε ασφαλιστικέ επιχειρήσει να έχουν τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα από τις δοκιμές αντοχής στις οποίες συμμετείχαν. Η διαδικασία σχετική θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να γενικευθεί αυτό και στις υπόλοιπες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν το έχουν πράξει. Περνάω τώρα στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασής μου. Κυρία Πρόεδρε, σπάνια το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι αναφερόμαστε σε καθήκοντα εποπτικά και έχουμε εδώ πέρα 20 μόνο εργαζόμενους στην ΕΙΟΠΑ, ένα 14 μόνο της 100 καταλαβαίνετε ότι αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μηδενική υποστήριξη. Αν πραγματικά θέλουμε μια πανευρωπαϊκή εποπτεία από την ΕΙΟΠΑ, θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις στον οργανισμό αυτό. Και προφανώς θα πρέπει να έχει και την κατάλληλη διακυβέρνηση η ΕΙΟΠΑ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να επενδύσουμε περισσότερο στο προσωπικό. Θέλουμε από την κατάρτιση πολιτικής να περάσουμε περισσότερο στην κατάλληλη εποπτεία και νομίζω ότι την άγουσα αυτή θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αυτά είναι τα βασικά μας συμπεράσματα. Προφανώς θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια της Επιτροπής σας για το ζήτημα αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επιστέλθουμε μαζί της και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό την παρουσίασή μου και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, τόσο σημαντική έκθεση. Είναι πρώτη έκθεση ελέγχου για την ΑΙΟΠΑ ε, και ως εκ τούτου είναι Βεβαίως όλες οι εκθέσεις σημαντικές, αλλά αυτή είναι πολύ σημαντική. Κύριε Κάρνμπαχ ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και μέσω αυτού το ελεγκτικό συνέδριο. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν επίσης ότι πρώτα απ' όλα ασχολούμαι με τους οργανισμούς, ε, κυρίως ε, στο γεωργικό τομέα. Αυτά όμως όλα άπτονται και των ασφαλιών. Ε, θα έλεγα λοιπόν να ασχοληθούμε πραγματικά με το θέμα αυτό, γιατί πάρα πολλοί και εδώ στο Κοινοβούλιο δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος σε αυτό τον τομέα. Εδώ ε, διακυβεύεται το μέλλον μας ε, παρά την οικονομική κρίση. Ε, θα τολμούσα να πω ευτυχώς σε πάρα πολλούς τομείς υπάρχει ακόμα εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά τα συστήματα ασφαλιών λειτουργούν και το θέμα της ασφάλειας ζωής. Ε, προετοιμάζοντας λοιπόν τη δουλειά μας για το μέλλον, θα ήθελα να θίξω δύο θέματα ε, που θίξατε κι εσείς. Το ένα είναι, αφορά το προσωπικό. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν σωστό να μας πει η Επιτροπή πώς προτίθεται να εξετάσει ε, το θέμα του προσωπικού πώς θα λυθεί το θέμα αυτό. Ακούσαμε 20 ε, συνεργάτες είναι μόνο το 14% των πόρων για το προσωπικό. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Ε, θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν κάποιες ανακατανομές σε επίπεδο προσωπικού πάντα όσον αφορά την ΕΟΠΑ ή μήπως, εγώ έτσι τουλάχιστον πιστεύω, χρειαζόμαστε επιπρόσθετο προσωπικό. Μετά, Κάτι άλλο. Ε, το είπατε πολύ κομψά, το δικαίωμα, το ε, πολύ ε, επιφυλακτικό δικαίωμα να ζητήσει κανείς πληροφορίες. Δειλά. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές ή από την έκθεση. Ε, φαίνεται επίσης ότι ε, σε πολλές περιπτώσεις δεν τους προσφέρεται η απαραίτητη υποστήριξη. Οι εθνικές αρχές ε, έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους σε πολλά επίπεδα και αυτό λοιπόν είναι καθοριστική σημασία και για το πώς ακριβώς ε, μπορεί να ε, ασκεί τι ε, εξουσίε τη και η ΟΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να δώσουμε πολλέ αρμοδιότητε στι εθνικέ αρχέ. Εσεί πώ πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και σήμερα στην ομιλία σα μιλήσετε επανειλημμένα για τη βελτίωση των νομικών διατάξεων. Μπορώ να κρίνω και να ερμηνεύσω από αυτό ότι ε, δεν θα πρέπει να είμαστε μόνο αυστηροί στην ερμηνεία των νομικών διατάξεων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαζόμαστε μία εκ νέου διατύπωση όλων αυτών των νομικών διατάξεων τι είδους διατάξεις χρειαζόμαστε έτσι ώστε και στο μέλλον να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία. Αυτή ήταν έτσι μια πρώτη προσέγγιση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη ε, δυνατότητα ε, να συζητήσουμε το θέμα. Θέλω να καλωσορίσω και να χαιρετήσω την κυρία Μπερέ στα γαλλικά, μέλο τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Έχουν προσκληθεί όλα τα μέλη τη για τη συζήτηση αυτή από τη, τη Γενική Διεύθυνση ε, Φίσμα ε, από τη Γενική Επιτροπή, ο κύριος Ράιεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Και φυσικά ε, δεν εκπροσωπώ την ίδια την ΕΙΟΠΑ, αλλά την ε- Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή όμως πολλές από τις ερωτήσεις αφορούν το ευρύτερο νομικό και νομοθετικό πλαίσιο για τη δραστηριότητα της ΕΙΟΠΑ, μπορώ να απαντήσω και σε αυτά ένα εισαγωγικό σχόλιο θέλω να προεξοφλήσω. Να μην λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων δεν είναι μόνο αρμόδια για τις ασφαλίσεις, αλλά και για τις επαγγελματικές συντάξεις. Και είναι πολύ σημαντική η πτυχή των ασφαλίσεων, αλλά εξίσου σημαντική που καλύπτει και πάρα πολλούς πόρους είναι και η διάσταση των επαγγελματικών συντάξεων. Ποιοι είναι οι πόροι. 112 υπαλλήλους έχει από το καταστατικό της, αλλά έχει και συμβασιούχους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες που φτάνουν συνολικά στους 150 και το ε, μοιράζονται αυτό οι ασφαλίσεις και οι συντάξεις. Ε, και τρεις μεγάλοι είναι οι τομείς δραστηριοτήτων. Το ένα είναι η ανάπτυξη ε, πολιτικής, δηλαδή συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Μελλοντική Νομοθεσία. Το δεύτερο είναι ο εποπτικός τομέας που ακούσατε ότι έχει 20 υπαλλήλου. και το τρίτο είναι ο τομέας οικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και αυτό αφορά τις εκθέσεις και τις ε, δοκιμές αντοχής, τα stress tests. Αυτά δεν τα κάνουν οι 20 υπάλληλοι που άκουσατε προηγουμένως, αλλά άλλοι επιπλέον που ασχολούνται με την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες ε, της ΑΙΟΠΑ. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου κάνει λόγο για ε, την αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των εποπτικών αρχών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2017 και ακόμα συζητούν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σωστά υπογραμμίζει ότι η πρόταση εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποπειράθηκε να λύσει μερικά από τα ζητήματα μόνο ε, που ε, μας απασχολούν σήμερα. Παράδειγμα, προτείνει κάποιες ενισχύσεις των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων ε, της ΑΕΟΠΑ για τα εσωτερικά μοντέλα, όχι να είναι ο βασικός ελεγκτής και επόπτης, αλλά να έχει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, στη διάθεσή της. Επίσης να έχει την εξουσία να γνωμοδοτεί προς τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές σε περίπτωση αποκλίνουσων ε, ερμηνεών των εσωτερικών μοντέλων για να υπάρχουν συνακτικά αποτελέσματα. Τώρα, για τις ε, δοκιμές αντοχής, τα περίφημα stress test. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, ε, πρότασή της ευθυγραμμίζει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής με την ΕΙΟΠΑ. Η EBA έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει ορισμένα μεμονωμένα στοιχεία από τις δικές αρμοδιότητες και αποτελέσματα μελετών και stress test. Η ΕΙΟΠΑ δεν το έχει ακόμα αυτό το δικαίωμα και θα το αποκτήσει με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω επίση να σα επιστήσω την προσοχή στο γεγονό ότι η πρόταση τη Κομισιόν συνοδεύεται και από ένα, μια νομοθετική οικονομική δημοσιονομική δήλωση που, αν εγκριθεί, θα σημάνει σημαντική αύξηση ε, στο προσωπικό της ΕΙΟΠΑ. Άρα αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα αυτό του προσωπικού. Και μια που είμαστε στο προσωπικό, αυτό είναι εκτός των ασφαλίσεων, είναι στις συντάξεις. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την πολιτική συμφωνία ε, στο τριμερή διάλογο συμφώνησαν το Δεκέμβριο για ένα νέο ε, συνταξιδοτικό προϊόν πανευρωπαϊκό. Εκεί θα γίνουν λοιπόν ε, αυτές οι ρυθμίσεις και ε, εκτός ε, τώρα της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών θέλω να αναφερθώ στις πολλαπλές ασφαλίσεις. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρθηκε σε διασυνοριακή δραστηριότητα και είναι γεγονός ότι στον τομέα αυτό υπήρξαν κάποιες ε, ασφαλίσεις, ε, κάποιοι φορείς ασφαλιστικοί οι οποίοι χρεοκόπησαν. για ε, ασφαλίσεις αυτοκινήτων, οχημάτων. Όταν χρεοκοπήσει, ας πούμε, μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει διασυνοριακές δραστηριότητες και παρουσία στην ασφάλιση οχημάτων, ε, θα πρέπει αυτό το θέμα να ρυθμίζεται. Βέβαια μετά τη διαδικασία της χειροκοπίας της αφαιρεγγιότητας. Ε, όχι όλα αυτά που έχουν να κάνουν μέχρι να κηρυχθεί η αφαιρέγγεια. Εκεί χρειάζεται βέβαια συντονισμός αλλά και περιορίζεται πάντα στην ασφάλιση των αυτοκινήτων και των οχημάτων. Βολιδοσκοπεί τον κλάδο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς αρχίζοντας από το συγκεκριμένο κλάδο ασφαλίσεων οχημάτων. Ε, αρμόδια επί τη ουσία ε, επιτροπή εδώ είναι η Επιτροπή ε, Ίντα. Για να δούμε μετά ε, τι γίνεται με την εκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σε διασυνοριακή βάση είναι δοκιμαστική, ας πούμε, πιλωτική αυτή η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ασφάλειες των οχημάτων. Και ένα τελευταίο είναι το Solvency ε, 2, το Φερεγκιότητα 2, που είναι το πλαίσιο που διέπει ε, την φερεγκιότητα των ασφαλίσεων. Και έχει εκεί τις περισσότερες διατάξεις και αρμοδιότητες και εξουσίες της ΕΙΟΠΑ. Είναι κάτι σχετικά νέο. Εφαρμόζεται την τελευταία τριετία. Επίκειται και έχει προγραμματιστεί για το 2020 μια μεγάλη αναθεώρηση ε, και έχουμε αρχίσει να την προετοιμάζουμε με διάφορες μελέτες ε, αντικτύπου. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και για αυτό το σκοπό και είναι πιθανό στα τέλη του 2020 να έρθει άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ε, τροποποίηση στην ε, σημερινή διαδικασία και το καθεστώς ε, Solvency 2. Και βεβαίως προσβλέπουμε στη συνεργασία του Κοινοβουλίου για αυτή την με πολύ μεγάλη αναθεώρηση το 2020. Θα περιορίσω εδώ τα σχόλιά μου. Με χαρά να σας απαντήσω αν έχετε ειδικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερές. Ευχαριστώ που καλέσατε τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων γιατί νομίζω ε, ότι θα ήταν χρήσιμο να έχετε και την άλλη θεώρηση και ε, ε, όψη των Μιλώ δε και ως συνεισηγήτρια που είμαι με τον Ότμαρ Κάρας για την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, ιδιαίτερα της ΕΙΟΠΑ. Ζητώ συγγνώμη από τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου για την καθυστερημένη άφηξή μου. Ε, είδα μόνο το PowerPoint, αλλά ε, νομίζω ότι έχω καταλάβει το πνεύμα σε γενικές γραμμές και περιμένω και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, για δύο θέματα θα ήθελα να μιλήσω εγώ ε, κατά κύριο λόγο. Το πρώτο έχει να κάνει με τα εσωτερικά μοντέλα. Διότι στην ΕΚΟΝ έχουμε μόνιμο καημό τη μείωση του κινδύνου ή τον επιμερισμό του κινδύνου. Ε, στον τραπεζικό τομέα έχουμε προχωρήσει πολύ προς την κατεύθυνση αυτή. Για τις ασφάλειες ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα των εσωτερικών μοντέλων είναι ευαίσθητο. Τώρα μπορεί κανείς να πει ε, το εσωτερικό μοντέλο το γνωρίζει καλύτερα η Εθνική Εποπτική Αρχή εκάστοτε. Θα μπορούσε επίσης όμως κανείς να ισχυριστεί ότι εκείνος που το γνωρίζει καλύτερα είναι ο πιο απρόθυμος ε, να βγει και να μιλήσει ξεκάθαρα και ειλικρινά όταν υπάρξει πρόβλημα. Εξού και η συστολή ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση ε, των εποπτικών ελέγχων και των εσωτερικών ελέγχων. Δεύτερος λόγος τι είδαμε στο τραπεζικό τομέα. Αυτό που είδαμε εκεί θα μπορούσε να επαναληφθεί ε, στον ασφαλιστικό κλάδο. Οι Αμερικανοί ε, που περιμένοντας τον Brexit είναι οι βασικοί μας ανταγωνιστές σε αυτά τα θέματα τα τραπεζικά και τα ασφαλιστικά. Ε, είδαμε τι έκαναν στον τραπεζικό τομέα με την Επιτροπή της Βασιλείας έχουν εξαπολύσει ανοιχτό πόλεμο κατά των εσωτερικών μοντέλων γιατί δεν έχουν αυτή την νομοθεσία. Ε, οι τράπεζες ακολουθούν μόνο στάνταρ, τυποποιημένες φόρμουλες. Και στην Επιτροπή της Βασιλείας ε, δυσκολεύονται πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά κράτη να υπερασπιστούν αυτά τα εσωτερικά μοντέλα. Λοιπόν, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και στις ασφάλειες. Διότι οι Αμερικανοί στην Επιτροπή της Βασιλείας χτίζουν διάφορες δομές όπου το θέμα της διεθνούς ρύθμισης του ασφαλιστικού κλάδου ε, θα τεθεί. Και αυτό που δεν κατάφεραν να περάσουν στις διμερείς ε, συνομιλίες για τη φερεγγιότητα 2 ε, οι Αμερικανοί θα το πετύχουν σε αυτό το διεθνές φόρουμ. Και υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ε, κάθε συμφέρον να διατηρήσουν το εσωτερικό μοντέλο γιατί καταλαβαίνουν τι γίνεται με την οικονομία της κάθε επιχείρησης και πώς λειτουργεί αυτή. Αλλά ε, θα ήταν καλύτερο αυτό να οργανωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν υπήρχε ευρωπαϊκή πραγματογνωμοσύνη για αυτά τα, ευρωπαϊκά, τα ιστορικά μοντέλα και έτσι αυτό θα εδραίωνε και την αξιοπιστία τους και ε, την ε, αποτελεσματικότητά τους και την αποδοτικότητά τους. Άλλο θέμα για τα εσωτερικά μοντέλα. Στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά είναι σωστό ο καθένα εφόσον τηρεί τις ε, προποθέσει, πληρεί μάλλον τις προϋποθέσεις, να μπορεί να χρησιμοποιεί τα εσωτερικά μοντέλα. Αλλά όταν έχει μια χώρα μικρή, με μια μικρή εποπτική αρχή, και τώρα δεν θέλω να ε, θίξω κανέναν λέγοντας μικρή χώρα, αλλά η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις εσωτερικό μοντέλο είναι κάπως περιορισμένη. και μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία σε μια μικρή ασφα... Ε, χώρα μπορεί να βασιστεί στην ευρωπαϊκή εμπειρία για να αναπτύξει το μοντέλο της. Δυστυχώς, και αυτό μου φάνηκε σωστό εμένα, δυστυχώς το Συμβούλιο η συνεσταλμένη κατά τα άλλα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν θέλει να ελέγχει η ίδια το εσωτερικό μοντέλο η ΕΙΟΠΑ όπως εγώ το προτείνω στις τροπολογίες μου απλώς ε, συντονισμό ζητάει και μια έτσι κάπως πιο οριζόντια ματιά. Αυτό έχει γνωρίσει θύελα αντιδράσεων στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε ε, στο Συμβούλιο για τη χρησιμότητά σας, για να μην μακρηγορώ, τι γίνεται με τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Ξέρετε ότι στις ασφάλειες η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών οδήγησε ε, σε τεράστιες υπερβολές και εξα... Ε, εξαμβλώματα με εταιρείε ταχυδρομικέ σειρίδες μαϊμού που πουλάνε ασφάλειες από χώρε που δεν έχουν ούτε την επιφάνεια ούτε την απαραίτητη αγορά για να υποστηρίξουν αυτά τα προϊόντα. Αλλά χρησιμοποιούν την ε, πνοευνοϊκή νομοθεσία για να ε, παίζουν σε ένα dumping νομοθετικό και δεν καθόλου τα δικαιώματα των καταναλωτών στις χώρες όπου πουλούν αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα. Και γνωρίσαμε πάρα πολλά σκάνδαλα τέτοιου τύπου τα οποία σήμερα ε, εξετάζει και ελέγχει η ΕΟΠΑ. Και όπου καμιά φορά η ΕΟΠΑ στερείται ε, δυνατοτήτων για να δώσει λύσεις και να μεσολαβήσει σε αυτές τις ε, περιπτώσεις. Μαζί με τον Ότμαρ Κάρας, λοιπόν, το συνεισηγητή μου, θα κάνουμε κάποιες προτάσεις χωρίς να περιορίζεται φυσικά η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αλλά να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η πραγματική αγορά της χώρας στην οποία πολλούν και διανέμουν αυτά τα προϊόντα, τα ασφαλιστικά. Χαίρομαι που είμαι εδώ και με χαρά θα περιμένω και τις εκθέσεις σας. Ευχαριστώ. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Ε, θα, θα μιλήσει ο Ράιν. μιλήσω στα γαλλικά για να απαντήσω στην κυρία Μπερές. Όσον αφορά τα εσωτερικά μοντέλα, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του Συμβουλίου για λόγους τυπικούς και πρωτοκόλου. Πάντως καταγράφω τα όσα υπόθηκαν όσον αφορά την εξέλιξη της συζήτησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και όντω αληθεύει ότι στα πλαίσια των διεθνών, του Διεθνούς Οργανισμού για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις International Association of Insurance Supervisors, ο Διεθνής Οργανισμός ε, Διεθνών Εποπτών για την ε, Ασφάλεια, προβλέπεται ότι όντως θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο προβλέπεται από την Επιτροπή της Βασιλείας για τις Ασφάλειες. Και επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη είναι υπέρ των συζητήσεων που γίνονται για τα ιστορικά μοντέλα στα διάφορα διεθνή φόρα και προσπιζόμαστε ιστορικά μοντέλα στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Καταγράφουμε λοιπόν όλε αυτέ τι παρατηρήσει. Όσον αφορά τώρα τι διασυνοριακέ δραστηριότητε, Συντοπίζουμε ότι υπάρχουν εδώ πέρα κάποιε υπερβολέ. Όντω, είχαμε περιπτώσει ασφαλιστικών επιχειρήσεων που χρεοκόπησαν, αλλά κυρίως τα φαινόμενα αυτά το είχα, τα είχαμε στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτων. Εκεί είχαμε τα πιο σημαντικά προβλήματα, εκεί είδαμε τις πιο σημαντικές υπερβολές και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τον τομέα αυτό για την πρώτη πρόταση που κάναμε σε μια απόπειρα ρύθμισης των κειμένων. Αν όλα ευοδοθούν και αν η πρόταση αυτή τελικά εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τότε σε ένα δεύτερο στάδιο θα δούμε αν θα καταφέρουμε να διευρύνουμε τον μηχανισμό αυτό και σε άλλους κλάδους ασφάλισης πέρα από τα αυτοκίνητα. Ξεκινάμε από τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων ως μια πρώτη απόπειρα ρύθμισης του προβλήματος αυτού. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα διάφορα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ότι ε, τοποθετήθηκαν στην κατεύθυνση που επιθυμούμε. Οι επιθεωρητές όταν ε, έλεγξαν τη δουλειά της ΕΟΠΑ σε αυτόν τον τομέα, κοιτάξτε, η δική μας η προσέγγιση είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς θεωρούμε δεδομένο οτιδήποτε ε, γράφεται ε, στη Λευκή Βίβλο από τους ε, νομοθέτες. Ε, υπάρχει βεβαίω το Solvency 2 και εμεί προσπαθούμε να αναλύσουμε πώ ακριβώ λειτουργούν όλα αυτά. Εδώ, επαναλαμβάνω βέβαια, τα έχω ξαναπεί, καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει σωστή κατανομή κινήτρων για όλου του παίκτε ε, για να ξέρουν και αυτοί πώ θα συμπεριφερθούν. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα τη εφαρμογή ε, του κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. Και βεβαίω, εδώ απαντώ στην κυρία Κάτμιν, πράγματι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και διαβάσαμε τις προτάσεις της Επιτροπής ε, αλλά αυτό δεν ήταν το δικό μας το καθήκον, δεν είναι δική μας δουλειά να τα εξτάσουμε λεπτομερώς. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι σε αυτές τις προτάσεις και σε κάποιες ε, τροπολογίες ε, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση προς το να αποκτάει η ΕΟΠΑ περισσότερες αρμοδιότητες για να έχει πληροφορίες που χρειάζεται. Η πρόσβαση στην ενημέρωση και η ανεξαρτησία της ΕΟΠΑ, αυτά τα δύο πράγματα από κοινού, νομίζω ότι θα λύνανε πολλά προβλήματα. Όχι όλα, αρκετά. Η ανεξαρτησία της ΕΙΟΠΑ σημαίνει περισσότερα δικαιώματα και ανεξάρτητες ε, εξουσίες, αρμοδιότητες. Και αυτό βέβαια είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το ξανασκεφτούμε και πρέπει να παγιωθεί στην ενωσιακή νομοθεσία. Σας καλούμε να τα σκεφτείτε όλα αυτά γιατί εμείς ε, βλέποντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα ε, και το κείμενο, το σώμα της νομοθεσίας βλέπουμε ότι αυτά διασυνοριακά δεν ένα πολύ καλό παράδειγμα ανέφερε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Εκεί έχουμε σαφώ κοινή αγορά. Τα αυτοκίνητα μετακινούνται σε ολόκληρο τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα. Υπάρχει εθνική ασφάλεια διασυνοριακή, ισχύει και διασυνοριακά. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε αυτόν τον τομέα, γιατί αλλιώς αυτό μπορεί να μας φέρει πολλά προβλήματα σε απλούς ανθρώπους, οι οποίοι οδηγούν τα αυτοκίνητά τους. Και Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι και πλούσιοι και φτωχοί. Οδηγούν όλοι αυτοκίνητο. Και αυτό είναι ένα ε, ξεκάθαρο παράδειγμα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Για άλλη λοιπόν μια φορά σας ευχαριστούμε που τοποθετηθήκατε ενεργά, που δεχτήκατε τη δική μας την έκκληση για δραστηριοποίηση και περιμένουμε, προσβλέπουμε στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και για να κλείσουμε κυρία Κάτμπαχ. Απλά ένα θερμό ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ε, ακούσαμε και προτάσεις από την κυρία Περές και νομίζω ότι ορισμένες από αυτές τις προτάσεις θα τις συμπεριλάβουμε στην τοποθέτησή μας. Πολύ ωραία. Πάει και αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης, το 8. Ε, και πάμε τώρα στο σημείο υπερθμών 9. Πανοραμική επισκόπηση για τις μεταφορές. Ε, ο κύριος Μπάλκο είναι ο εισηγητής ε, και ε, ο κύριος Τσέλερ θα αντικαταστήσει την ε, κυρία Σμιτ. Ο κύριος Μπάλκο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καλησπέρα σας λοιπόν κυρία Πρόεδρε, κυρία Συγήτρια, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πανοραμική επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σχετικέ προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι μεταφορέ, όπω ξέρουμε, επηρεάζουν την καθημερινή ζωή πολλών πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα στρατηγικό τομέα για την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπηρεσίε του τομέα των μεταφορών αντιστοιχούν περίπου σε 11 εκατομμύρια θέσει απασχόληση. Οι μεταφορέ είναι ακρογωνιαίο λίθο τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα ορθά σχεδιασμένα βιώσιμα πολυτροπικά δίκτυα μεταφορών είναι πολύ σημαντικά για τη σωστή ορθή λειτουργία της ευρωπαϊκής Ιστορικής αγοράς. Οι αποτελεσματικές μεταφορικές υπηρεσίες και σχετικές υποδομές, όμως, θα πρέπει να εκμεταλλεύονται και τι τα οικονομικά προτερήματα μάλλον των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η προστιθέμενη αξία της πανοραμικής αυτής επισκόπησης, όπως και οι προηγούμενες επισκοπήσεις που έκανε στον τομέα αυτό το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο παρέχουν μια αναλυτική περιγραφική επισκόπηση του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα συγκεκριμένο τομέα, εν προκειμένου στον τομέα των μεταφορών δίνοντας προσβάσιμε και ξεκάθαρε πληροφορίε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουμε ως στόχο να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις δράσεις στον τομέα των μεταφορών, να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονομένα κράτη-μέλη προκειμένου να πετύχουν τους στόχους στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπω το είπαμε, οι μεταφορέ αποτελούν τομέα συντρέχουσα αρμοδιότητα μεταξύ των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η ευθύνη για την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των μεταφορικών υποδομών βαρύνει κυρίω στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει κυρίω ω καταλήτη μέσω τη χρηματοδότηση τη για να καλυφθούν συγκεκριμένε ανάγκε. Στην πανοραμική λοιπόν αυτή επισκόπηση επικεντρωνόμαστε στις επενδύσεις πρέπει να γίνουν στον τομέα των υποδομών, καθώς επίση και σε κάποια οριζόντια θέματα, τα οποία εντοπίσαμε σε 13 πρόσφατους ελέγχους που κάναμε στους πέντε βασικούς τρόπους μεταφοράς, δηλαδή σοδικές, διαδρομικέ, αεροπορικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές βάσει των συστάσεων που γίνονται στους ελέγχους αυτούς, αλλά και βάσει υπορισμάτων και συστάσεων άλλων ελέγχων και ερευνών που έχουν γίνει από άλλους οργανισμούς, καταλήγουμε σε μια οριζόντια ανάλυση των βασικών προκλήσεων και των γενικότερων τάσεων που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των μέτρων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανοραμική αυτή επισκόπηση απαρτίζεται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρέχει μια σφαιρική παρουσίαση των βασικών πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το μέτρο μεταφορών. Αναφέρεται στην, στο υποκείμενο πλαίσιο διακυβέρνηση καθώς επίσης και στη χρηματοδότηση. Το δεύτερο τμήμα της επισκόπησης αυτής αναφέρεται στην τρέχουσα κατάσταση και στους βασικούς τομείς όσον αφορά το μέτρο μεταφορών, ενώ το τρίτο τμήμα αναφέρεται στα οριζόντια ζητήματα και κυρίως στις βασικές προκλήσεις. Καθότι πιέζει ο χρόνος, εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στο δεύτερο και τρίτο τμήμα Τη επισκόπηση αυτή. Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τι αναδυόμενε τάσει στον τομέα των μεταφορών, μπορούμε να πούμε ότι ο όγκο των μεταφορών κατά σταθερό τρόπο αυξάνεται και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τόσο για τι επιβατηγές όσο και τι εμπορευματικέ μεταφορέ. Η αύξηση στον όγκο των μεταφορών μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένε προκλήσει όσον αφορά συγκεκριμένου τομεί μεταφορών και ήδη μπορούμε να πούμε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική και οικονομική ανησυχία, η οποία στοιχίζει αυτή τη στιγμή 140 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε έτος. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν τον πρωταρχικό τρόπο μεταφορών για τους επιβάτες και για τους αγαθές και για τα αγαθά, με συγχωρείτε. Επικεντρωνόμαστε στην έκθεσή μα στι εγχώριε μεταφορέ, δηλαδή αφήνουμε εκτό τι θαλάσσιε και νέε μεταφορέ και εκεί συνειδητοποιούμε ότι η μεταφορά μέσω αυτοκινήτου αντιστοιχεί στο 83% τη γενικότερη μεταφορική δραστηριότητα όπως αυτή εκφράζεται σε επιβατοχιλιόμετρα. Όσον αφορά τι μεταφορέ εμπορευμάτων, έχουμε ένα στόχο 30% μετατόπιση δηλαδή των αγαθών αυτών από τι οδικέ μεταφορέ προ τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ, Ο στόχος αυτός γίνεται 50% με χρονικό ορίζοντα το 2050, γιατί θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε πιο φιλοπεριβαλλοντικέ μορφέ μεταφορών. Μπορούμε πάντω να πούμε ότι όσον αφορά τον μερίδιο οδικών μεταφορών για την εσωτερική μεταφορά εμπορευμάτων έχουμε μια αύξηση 75,1% το 2011 όσον αφορά τις συνολικές μεταφορές, ποσοστό που έχει γίνει 76,4% το 2016. Το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια ειδική έκθεση όσον αφορά τι σιδηροδρομικέ εμπορευματικέ μεταφορέ, την οποία σα παρουσίασα στην Επιτροπή αυτή στο παρελθόν και είχαμε και πέρα από την παρουσίαση αυτή στην Επιτροπή σας και σε μια άλλη Επιτροπή πολύ σημαντικές συναντήσεις και συζητήσεις με άλλα διαφερόμενα μέρη κατά τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής. Συγκρίναμε στην έκθεση αυτή τις βασικές προκλήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις οδικές, επιβατικές και τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καθώς επίσης και τις βασικές προκλήσεις που έχουμε στη μετατόπιση της Μεταφορά εμπορευμάτων από τι οδικέ σε άλλε μεταφορέ. Α μην ξεχνάμε ότι ενώ ο στόχο αυτό ακόμα δεν έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν άλλε χώρε όπω η Αυστραλία, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν καταφέρει να πετύχουν το στόχο αυτό, φτάνοντα μάλιστα σε ένα 40%. Α μην ξεχνάμε επίση ότι οι μεταφορέ έχουν αρνητικέ εξωτερικέ συνέπειε όπω τροχιά ατυχήματα, εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, τον σφαιρική ρήπανση, χορύπανση. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα κοινωνικό και οικονομικό κόστος, όπως είχαμε πει και στην ειδική έκθεση 19 κάθος 2018, αναφερόμενοι τότε στις, στους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, προσπαθήσαμε να δούμε στην περίπτωση αυτή πώς τα συστήματα τελών τα οποία εφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν τελικά να συνδυάσουν δύο βασικές αρχές. Την αρχή ο χρήστης πληρώνει και την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μα απασχόλησε είναι πολυτροπικό, πολυτροπικότητα. Η πολυτροπικότητα ουσιαστικά αναφέρεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών διαφορετικών μέσων μεταφορά στα πλαίσια τη ίδια διαδρομή του ίδιου ταξιδιού και αυτό αποτελεί στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε μέσω τη πολυτροπικότητα να πετύχουμε την αλλαγή του τρόπου εκτέλεση των μεταφορών, το λεγόμενο modal shift, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι πολυτροπικές μεταφορές δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αναφερόμαστε στην έκθεση αυτή και στα ευφυή συστήματα διαχείριση των μεταφορών που έχουν να κάνουν με διάφορου τρόπου μεταφορών. Εδώ πέρα έχουμε κάποια αρμόδια συστήματα όπω το ERTMS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα διαχείριση τη Σιδηροδρομικής κυκλοφορία, για το οποίο μάλιστα είχαμε και μια ειδική έκθεση, την υπαριθμών 13 2017. Έχουμε επίση και ένα άλλο πρόγραμμα, το CESAR, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, ειδική έκθεση για τον οποίο σα παρουσίασε άλλο συναδελφό μου στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι η επιτυχή συντονισμένη ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να πετύχουμε ένα πανευρωπαϊκό, πολυτροπικό και πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί, έχουν διατεθεί στα πλαίσια του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής από το 2000, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2020, ενώ επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται στα πλαίσια του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη μέχρι τα τέλη του 2017. Μετά την οικονομική κρίση του 2008 μειώθηκαν οι επενδύσεις στις ε, υποδομές μεταφορών. Προκειμένου όμω να καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε σημαντικού χρηματοδοτικού πόρου. καθότι τα δημο, οι δημόσιοι πόροι πλέον οι δημόσιοι πόροι είναι περιορισμένοι, επενδύουμε όλο και περισσότερο στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των υποδομών μεταφορών. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πορίσματα τη ειδική μα έκθεση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα διαχείριση τη Ιδρονομική κυκλοφορία. ERT TMS. Μολονότι είχαμε ήδη σημαντική συμβολή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και την προσφασιμότητα, περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η βασική ευθύνη για την κατασκευή υποδομών επιβαρύνει κυρίω τα κράτη-μέλη. Παράλληλα όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει τα λεγόμενα κριτήρια του Μάστρικ όσον αφορά το ποσοστό του δημοσίου χρέους ως προς το εθνικό ΕΠ. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια πολλές φορές σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε σχέση με την ικανότητα επενδύσεων των κρατών μελών σε συγκεκριμένες υποδομές μεταφορών οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να δούμε πώ μπορούμε να συσχετίσουμε αυτού του δύο αντιτιθέμενου στόχου. Μείωση του δημόσιου χρέου από τη μία πλευρά και αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε υποδομέ μεταφορών από την άλλη. Επίση, το ποσοστό ανάπτυξη συγκεκριμένων υποδομών αποτελεί αλλά παρουσιάζει στέρηση, ιδίω σε διάφορε ανατολικέ περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, τα κεντρικά δίκτυα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών έχουν ολοκληρωθεί ενώ υπολείπονται σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Πιο αργά, λέει η Πρόεδρος, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν και διερμηνήσει. Τα κεντρικά λοιπόν δίκτυα στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών έχουν ολοκληρωθεί, πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν σε ορισμένα κράτη-μέλη, ενώ υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία υπολείπονται πάρα πολύ στο στόχο αυτό. Έχουμε ακόμα κάποια απουσία συγκεκριμένων κυκλοφοριακών συνδέσμων, ενώ υπάρχουν ακόμα σημεία συμφόρηση σε πολλά μεταφορικά δίκτυα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω επιβαρύνονται εδώ πέρα τα σημεία διέλευση των συνόρων. Επίση, οι προπολογισμοί που προβλέπονται για τη συντήρηση των οδικών και μεταφορικών υποδομών δεν έχουν του απαραίτητου πόρου και επίση δεν ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες δημιουργίας υποδομών, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές ακόμα εκκρεμούσες υποχρεώσεις συντήρησης. Οι οδικέ μεταφορέ είναι αυτέ οι οποίε πιο γρήγορα κατάφεραν να προσαρμοστούν στι τροποποιήσει τη αλυσίδα διοικητική μέρημνα, καθώ επίση και στην, στις νέες, στα νέα γεωγραφικά εμπορικά μοντέλα τα οποία προέκυψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ βλέπουμε ότι οι άλλοι τρόποι μεταφορά και ιδίω οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ απαιτούν ακόμα περισσότερο χρόνο προκειμένου να καταφέρουν να ανταποκριθούν και προκειμένου να καταφέρουν να αρμονίσουν τα εσωτερικά του συστήματα διαχείριση κυκλοφορία. Επίση, υπάρχουν ακόμα κάποιοι στόχοι που πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε όσον αφορά το άνοιγμα τη αγορά και την ελεύθερη, ελευθέρωση των υπηρεσιών, ιδίω όσον αφορά τον σιδηροδρομικό τομέα και τον τομέα των αεροπαρικών μεταφορών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η ελευθέρωση τη αγορά σιδηροδρόμων έχει επιτευχθεί μόνο εν μέρη στα κράτη-μέλη, ενώ η εικόνα διαφέρει πάρα πολύ από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νεοεισερχόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στι συνδρομικέ υπηρεσίε, οι οποίε βλέπουμε ακόμα ότι την είναι πλήρου εκμετάλλευση από του ήδη κατεστημένου φορεί. Επίση, ο τομέα τη αγορά τη τέταρτη δέσμη σιδηροδρόμων θα θεραπεύσει την κατάσταση αυτή, ελπίζουμε ήδη από τον Ιούνιο του 2019. Βλέπουμε επίση ότι ο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και οι σχετικέ μεταφορέ παραμένουν αρκετά κατακαιρματισμένε. Επίση, ο τομέα των μεταφορών έχει και κάποιε ευρύτερε επιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί στο 1 τέταρτο των γενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί τελικά μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον στόχο που έχει θέσει για την εξάλληψη των ανθρακούχων εκπομπών, οι οποίες όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά από το 2014 και μετά άρχισαν και αυξάνονται. Οι οδικές μεταφορές είναι οι πλέον υπεύθυνε για τις εκπομπές αυτές, αντιστοιχούν στο 72% των συνολικών εκπομπών από το τομέα των μεταφορών για το 2016. Το 2017 το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο εξέδωσε μία πανοραμική επισκόπηση όσον αφορά την ενέργεια και την κλιματική κλιματική στην οποία έκθεση μεταξύ άλλων συμπεριλαμβανόταν μια σφαιρική επισκόπηση των ε, ελέγχων του τομέα μεταφορών έλεγχοι που έχουν γίνει από ανώτατα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που είχαν θέσει ως στόχο τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της μείωσης των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου και άλλο αντικείμενο του ελέγχου αυτού ήταν κατά πόσο το μέσο των μεταφορών είχε όντω εφαρμόσει συστήματα εξάλληψη των θρακούχων εκπομπών. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται να εξελίξει μία άλλη έρευνα που έχει να κάνει με τα ευφυή συστήματα διαχείριση μεταφορών, προκειμένου να καταλήξουμε σε πραγματικά πανευρωπαϊκά ευφυή συστήματα μεταφορών. Η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση, η από κοινού κινητικότητα είναι αναδυόμενε τάσει οι οποίε θα συμβάλλουν στο να γίνουν πιο αποδοτικέ οι μεταφορέ μα. Οι νέε όμω τεχνολογίε και τα νέα μοντέλα φέρνουν και νέε προκλήσει, ιδίω όσον αφορά την καταλληλότητα του νομοθετικού πλαισίου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητήματα ασφάλεια, ζητήματα λογοδοσία και ευθύνη και ζητήματα ασφάλεια δεδομένων. Περαιτέρω, η προσαρμογή των μεταφορικών υποδομών σε νέα μοντέλα κινητικότητας και η ανάπτυξη νέων υποδομών για καθαρές και για καθαρά και εναλλακτικά καύσιμα είναι νέες προκλήσεις για τις οποίες θα πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις. Διακόπτη η Πρόεδρος, μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ πολύ και πάλι σας τονίζω ότι διαβάζετε πολύ γρήγορα για τους διερμηνείς. Ολοκληρώνοντας, Μολονότι η πανοραμική αυτή επισκόπηση αναγνωρίσει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών και όσον αφορά το άνοιγμα τη εσωτερική αγορά μεταφορών και μολονότι αναγνωρίζεται ότι έχουν εγκριθεί κάποια μέτρα για την εξάλληψη των αθρακούχων εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών, υφίστανται έξι βασικέ προκλήσει, τι οποίε θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών. Πρώτον, αντιστοίχηση συναφών και εφικτών στόχων και προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταφορών με του διαθέσιμου πόρου. Δεύτερη πρόκληση, η θέσπιση αποτελεσματικών εργαλείων επιβολή τη νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσει των κρατών μελών ω προ υποδομέ ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δίδοντα ιδιαίτερη προσοχή στα διασνοριακά τμήματα και στα προβλήματα κυκλοφορικής συμφόρησης που παρουσιάζονται εκεί. Τρίτη πρόκληση είναι εστιάσουμε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προτεραιότητες με την υψηλότερη ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Τέταρτη πρόκληση. Η βελτίωση του προγραμματισμού, τη εφαρμογή και τη παρακολούθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέμπτη πρόκληση. Διασφάλιση τη επρακού συντήρηση και τη βιωσιμότητα των υποδομών. Και η τελευταία πρόκληση που έχουμε εντοπίσει είναι η ενίσχυση των προσπαθειών για τη μετατόπιση περισσότερων αγαθών σε άλλους τρόπους μεταφοράς εκτός των οδηγών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Τσέλα, εκ μέρους της ηγήτριας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπάλκο και τους ε, συνεργάτες του ε, του συνεργάτε του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αυτή την έκθεση. Έκθεση που αφορά στη βελτιστοποίηση ε, του τομέα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό που μα απασχολεί είναι οι προκλήσεις. Η γνωμοδότηση τη συναδέλφου είναι η εξή. Ευχαριστεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτή την εκτεταμένη ανάλυση των υποδομών που χρηματοδοτούνται από τον ενωσιακό προπολογισμό. Οι επενδύσει αυτέ αφορούν τους τα πέντε μέσα μεταφορά και και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς μια γενική εικόνα τη στιγμή που υπάρχουν μεμονωμένες εκθέσεις οι οποίες δίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία αλλά χάνεται κάπου ε, το δάσος. Ε, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι το εξής. Η επέκταση των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει με διαφορετικό ρυθμό, όπου βέβαια όσον αφορά την ποιότητα και την διαθεσιμότητα των υποδομών, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ε, βελτίωσης κυρίως σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, σε ορισμένα κράτη έχουν προχωρήσει τα συστήματα, τα έχουν ολοκληρώσει, αλλά πάλι όμω έχουν ακόμα πάρα πολλά να κάνουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά ε, όπου ακούμε για αυτές τις διαφορές ανάμεσα σε κράτη. Θυμάμαι πολύ καλά μια άλλη ιδιαίτερη ειδική έκθεση της, του Ελληνικού Συνεδρίου που διαπίστωσε ακριβώ τα ίδια. Δεν θα επαναλάβω την περίληψη του του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά θα περιοριστώ σε δύο προτάσεις γιατί παρουσιάζουν τα προβλήματα με τον βέλτιστο τρόπο. Ε, και ρωτάει κυρία Σμίτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο σε αναλύσει ε, των μεταφορών διαπιστώνει πρώτον ότι οι κανόνε είναι πολύ περίπλοκοι και δεύτερον πρέπει να βελτιωθεί και μπορεί να βελτιωθεί ο σχεδιασμό. Πότε λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε βελτιώσει, γιατί έχω κουραστεί πια να ακούω συνεχώ τα ίδια, αλλά τελικά δεν είναι η απόψη εκείνη που θέλουμε να ακούσουμε. Η ε, Κομισιόν πώς μπορεί να εξασφαλίσει τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται με τον ε, καλύτερο δυνατό τρόπο τη στιγμή που μόνο τυχαία και σπορδικά γίνονται μελέτες σκοπιμότητας και κόστους-οφέλους επειδή, κυρία Σμιτ δηλαδή, είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, γνωρίζω τα προβλήματα όταν πρόκειται να μεταφερθούν οι μεταφορές από τις οδικές αρτηρίες στα τρένα. Όμως αυτά πολλές φορές είναι προβλήματα για τα οποία φταίνε τα ίδια τα κράτη-μέλη. Εγώ ε, έχω επιφυλάξει σε, όσον αφορά αυτά που λέει το ελεκτικό συνέδριο. Συνέδριο αναφέρεται σε κάποιες ε, ε, φορείς ειδικού συμφέροντος, αλλά θα έπρεπε να δώσει περισσότερο στα θέματα των φορολογουμένων. Ε, είχαμε και μία έκθεση που ανέφερε και ο κ. Μπάλκο ε, σχετικά με τις διαδρομές υψηλής ταχύτητας. Αυτό που ενδιαφέρει είναι οι διασυνοριακές διαδρομές να συνδυάζονται γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν ε, τα απαραίτητα κίνητρα. Το να επεκταθεί κανείς και άλλα 15-20 χιλιόμετρα πέρα από τα κίνητρα. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να σε εκπλήσει που εξακολουθούν να επεκτείνονται οι οδικές μεταφορές. Ε, μία ε, μεγάλη τρή, η DHL, μου είπε ότι το 60% των μεταφορών της ε, γίνονται αεροπορικά, το 40% με φορτηγά, με το τρένο καθόλου, γιατί δεν υπάρχει αρκετή ευελιξία. Η κυρία Σμιτ λοιπόν λέει σε αυτή την περίπτωση ότι ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να εξαφανιστεί εν τη γενέση του. Ε, πότε η Κομισιόν θα αλλάξει το μοντέλο που παρουσιάζει. Ε, θέλουμε τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα. Δεν συμβαίνει αυτό. Και πού οφείλεται αυτό, τη στιγμή που τα κράτη-μέλη παίρνουν τα κονδύλια, αλλά όταν πρόκειται να εφαρμόσουν προγράμματα σκέπτονται εθνικά και η συνάδελφος κυρία Σμιτ ευχαριστεί πολύ για ε, τις απαντήσεις που θα δοθούν. Και εγώ, ο κύριος Τσέλερ, λέω, ο υποφαινόμενος δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αξιολογεί τις προσπάθειες ε, που καταβάλλονται και εξωενωσιακοί ε, παράγοντες να παρεμβαίνουν στον προγραμματισμό μας. Παραδείγματο χάρη, στον δρόμο του μεταξιού, στη στρατηγική της Κίνα, ε, υπάρχουν ε, λιμάνια που ανήκουν σε Κινέζου σχεδόν ε, καθ' ολοκληρία, και τώρα προβλέπεται αυτό αυτή η διασύνδεση Βελιγραδίου-Βουδαπέστη, θα πράξουν και άλλες διασυνδέσεις, οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Όλα αυτά πώς εντάσσονται στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό που αν λάβουμε υπόψη μα την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα εμβαλωματικός, κυρίως όσον αφορά στην εφαρμογή. Ευχαριστώ. άλλο. Ε, κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μπάλκο για την εξαντλητική του έκθεση και παρουσίαση, πάρα πολύ χρήσιμη, πανοραμική και γενικά το ελεκτικό συνέδριο είναι πάρα πολύ ε, βοηθητική αυτή και πάντα ε, ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε ξανακούσει και δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα, συν τα καινούργια που έρχονται να προσθεθούν. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο το εξής. Δεν θέλω περιπτυσολογία και περιγραφή. Εντάξει, καλή είναι και αυτή, αλλά δεν μας δίνει το όραμα που θέλουμε εδώ, ε, ούτε τη θεώρηση που ζητούμε στην Επιτροπή μας, την εικόνα που θέλουμε να έχουμε. Αυτά που μας λέτε είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα για την Επιτροπή Μεταφορών, όχι για τούτη εδώ την Επιτροπή. Κύριε Πάλκο, το ελεγκτικό συνέδριο πώς αξιολογεί λοιπόν την ε, χρησιμότητα των κονδυλίων, δηλαδή πιάνουν τόπον. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι πολλά τα κονδύλια, οι διάφοροι πόροι και τα ταμεία ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τις υποδομές, για τις μεταφορές και για τις υπηρεσίες μεταφορών γιατί ε, ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ ε, θετικά ότι στις τελευταίες προκήρυξεις του διαγωνισμού του Connecting Europe, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τις υπηρεσίες, όχι μόνο για τις υποδομές. Ρωτώ λοιπόν, αυτά τα έχετε ιεραρχήσει, τα έχετε αξιολογήσει. Ε, ποιος τύπος χρηματοδότησης προσφέρεται καλύτερα. Γενικά γίνεται λόγο για επιδοτήσει, αλλά εδώ έχουμε πολλά ταμεία, τα διαρθωτικά ταμεία, το Ταμείο συνοχή, την διευκόλυνση συνδέοντα τη Ευρώπη. Ε, υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, όπω είναι και το σχέδιο Juncker, το ΕΦΣΥ. Λοιπόν, εσεί, τι πιστεύετε για όλα αυτά, για του διάφορου μηχανισμού χρηματοδότηση που υπάρχουν. Επίση ακούμε και λέτε κι εσεί και είναι και γεγονό ότι υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα με στενοπούς και δυσκολίες κυρίως στο σιδηρόδρομο που δεν είναι ούτε καν εθνικά ζητήματα αλλά είναι άλλη τάξη προβλήματα. Εσείς πώς αξιολογείτε εκεί ακριβώς την υλοποίηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεπερνάμε τα παραμεθόρια προβλήματα στο σιδηρόδρομο. και το κινέζικο, συνικό πρόβλημα εντό εισαγωγικών που ανέφερε ο κύριος Τσέλερ. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί πολύ συχνά, και όχι μόνο στι υποδομές, έρχονται οι Κινέζοι γιατί δεν έρχονται Ευρωπαίοι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το εργασιακό κόστος. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πατριωτισμός. Γιατί αν ο πατριωτισμός είναι υπερορθολογικός, για να μην πω τίποτα χειρότερο, θα μας τη φέρνουν κανονικά πάντα οι Κινέζοι. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ρόιτερς. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Μπάλκο, επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καλή χρονιά τώρα που αρχίζει το νέο έτος σε όλους στην Επιτροπή σας και εσείς προσωπικά και ήθε ε, οι εκθέσεις που συζητάτε εδώ και αποφασίζετε να είναι τόσο σημαντικές σε μια τόσο σημαντική χρονιά όπως είναι το 2019 που είναι και εκλογικό έτος. Και νομίζω ότι εδώ αντανακλώ και το αίσθημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η πανοραμική εικόνα είναι μια πάρα πολύ καλή επισκόπηση και μας δείχνει τι έχει κάνει το Ελεκτικό Συνέδριο τα τελευταία έτη ε, για τις μεταφορές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ ε, καλά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχει ο τομέας των μεταφορών. Και εμείς κάναμε προτάσεις και για μένα ε, η επιθυμία μου και ευχή μου θα ήταν να δώσει συνέχεια το Κοινοβούλιο ε, στις προτάσεις ε, που καταθέσαμε στις τρεις δέσμες μέτρων για την κινητικότητα και τις σημαντικές προτάσεις για τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτρέψτε μου να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες και να απαντήσω σε ερωτήσεις της κυρίας Σμιτ, του κυρίου Τσέλα και της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι εργαζόμαστε πολύ σκληρά για κάποιες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα ε, στις μεταφορές. Έτσι θα έχουμε μια κινητικότητα με λιγότερες εκπομπές. Όπως σας είπα έχουμε καταθέσει τρεις δέσμες, τρία πακέτα. Η Europe on the Move, μια κοινωνική ε, μετάβαση σε μια καθαρή συλλογική και μαζική μεταφορά για όλους και επίσης δέσμες που έχουν να κάνουν με τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και των καυσαερίων αλλά και με τη διευκόλυνση ε, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ε, τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τις συνδυασμένες μεταφορές. Για να σας αναφέρω επιγραμματικά μόνο λίγες από τις προτάσεις που έχουμε κάνει εδώ η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ υψηλή και έχει γίνει και πάρα πολύ κατανοητή και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά κάνουμε και προτάσεις ε, ε, για να οθήσουμε ε, σε επενδύσεις στις υποδομές. Μια πρόταση για ένα Connecting Europe Facility δεύτερης γενιάς που συνεχίζει την πολιτική του 2014 και μέχρι το 2030 θα έχουν δημιουργηθεί τα κεντρικά, το κεντρικό δίκτυο στις ε, μεταφορές, το διευρωπαϊκό. Ο κύριος Μπάλκο το είπε και αυτός ότι χρειάζεται χρόνο για να στηθεί το ERTMS ή το ΣΕΖΑ ως ενιαία ευρωπαϊκά συστήματα ή ε, να λυθούν τα ε, διασυνοριακά προβλήματα ή συμφορήσεις γιατί λείπουν κάποια χιλιόμετρα σιδηροδρόμου. Χρειάζονται δύο λοιπόν τέτοιες προγραμματικές περίοδοι για να υλοποιούνται σωστά όλα αυτά τα προγράμματα. Ακριβώς εδώ βρισκόμαστε μετά από τέσσερα χρόνια υλοποίηση, Τι διαπιστώνω. Είναι καλύτερη σήμερα η μετακίνησή μας κύριε Τσέλερ. Νομίζω ναι. Ε, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη για πρώτη φορά ε, έδωσε με κεντρικό τρόπο χρήματα ε, που τα έχει αφιερώσει απολύτως στα μέσα μεταφορών ε, που είναι υπέρ του περιβάλλοντος, σιδηρόδρομος, εσωτερικές πλωτές οδοί και όχι στην αεροπορία ούτε στις οδικές μεταφορές εκτός από θέματα ασφαλείας φυσικά. Και για πρώτη φορά έχουμε χρήματα εστιάσει στις χώρες συνοχής γιατί στο σημερινό ΣΕΦ υπάρχουν δύο φάκελοι. Ο ένας ε, ε, για όλα τα κράτη αλλά και ένας δεύτερος με κεντρική διαχείριση για τις χώρες συνοχής. Και πραγματικά έχει κάνει αυτό τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν γιατί επικεντρώνονται σε διασυνοριακά έργα αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Βαλτικές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Χρηματοδοτούμε εκεί όλα τα ε, προγράμματα ε, και τα έργα που είναι δύσκολα για εκείνα. Και ξέρετε ότι έχουμε την αρχή ε, το απορροφάσει το χάνεις, use it or lose it το κονδύλι. Ε, οπότε αν μείνουν αναπορόφητοι κάποιοι πόροι, ε, επιστρέφονται. Θα πρέπει λοιπόν τώρα ε, να δούμε και ένα τρόπο να δίνεται αυτό στις χώρες συνοχής με ένα είδος ανταγωνιστικού φακέλου, να κάνουν ένα διαγωνισμό μεταξύ τους, μια κούρσα οι χώρες της συνοχής. Αυτό είναι πολύ αμφισβητούμενο και αμφιλεγόμενο. Ε, αλλά ε, έχουμε κάνει ε, μεγάλο δρόμο, όπως το Rail Baltica που βγαίνουμε στη φάση της προκήρυξης διαγωνισμού. Θα χρειαστεί μέχρι το 2025-2026 η εκτέλεση αυτών των έργων κατά το διαγωνισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για την επόμενη περίοδο τι επόμενε πολιτικές δημοσιονομικέ προοπτικέ, και όταν έρθουμε με την, στην επόμενη πανεοραμική παρουσίαση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, δεν θέλουμε να ακούμε μόνο ότι το εξετάζουν αλλά ότι το υλοποιούν όταν θα έρθετε εσείς η κυρία Σμιτ να μας ζητήσετε το λόγο. Αυτό ακριβώς θέλουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό αποσκοπούμε. Αυτό συμπεριλαμβάνει και κάποια άλλα στοιχεία που ε, αναφέρατε για την επιλεξιμότητα και για τις πολυτροπικές, δηλαδή συνδυασμένες μεταφορές ή τη μεταφορά από τον αυτοκινητόδρομο στο σιδηρόδρομο. Ας ε, το, έχουμε συζητήσει, ας πούμε, το έργο στο Μπρένερ ή την υπερταχεία Μα ε, πώς θα το κάνουμε αυτό όταν ε, ε, είναι τόσα πολλά τα φορτηγά που περνούν τις Άλπεις. Μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά το, αυτό, η σύραγγα στον Πρένερο θα χρειαστεί μέχρι το 2027. Ε, πώς θα κάνουμε τη μετάβαση στο σίδηροδρόμο. Οι κινέζικες επενδύσεις είναι γεγονός βεβαίως. Ο Πειραιάς, ας πούμε, είναι στα χέρια της Κόσκο, των Κινέζων επενδυτών. Ε, αναφερθήκατε στη σιδηροδρομική σύνδεση Βελιγραδίου, Βου, δαπέστες. Αυτό τώρα είναι μια υπόσχεση εντό εισαγωγικών, γιατί μας τατάζουν μόνο, δεν έχουμε δει να υλοποιούνται. Υπάρχουν ε, οι αρμόδιες ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Επιτροπής, DG Budget, άλλε γενικέ διευθύνσει. δεν είμαστε καταρχήν ε, αντίθετοι με αυτέ τι επενδύσει, αλλά θα πρέπει να σέβονται το, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δίκαιο ανταγωνισμού, το δίκαιο διαγωνισμών, το περιβαλλοντικό δίκαιο κτλ. Όταν υπάρχει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή πραγματικά κινούμεθα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ε, των νέων αυτών πολιτικών με ε, τη διαδικασία και, πους και pull, δηλαδή ε, με επενδύσεις και με νομοθεσία. Έτσι ώστε όταν νομοθετούμε να ξέρουμε ότι υπάρχει και εναλλακτική λύση και δεν γίνονται όλα από, μέσω των οδικών μεταφορών ή των ε, αεροπορικών μεταφορών που τόσο ρηπαίνουν οι οδικές. Όπως αναφερθήκατε και εσείς στη DHL. Κυρία Γιάλα, μιλήσατε για τις κινέζικες εταιρείες. Βεβαίως χρειάζεται προσοχή. Και μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο κοιτούμε ε, ποια είναι η χρηματοδότηση και τι κάνει το ελεγκτικό συνέδριο και σε προηγούμενες εκθέσεις το έκανε, ε, έχει κάνει συστάσεις τις οποίες ακολουθούμε και αυτή η επισκόπηση, ε, η πανοραμική μας επιτρέπει θαυμάσια να το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Μπάλκο, αν έχει την καλοσύνη, με την πρέπουσα ε, διάρκεια παρακαλώ να κρατήσετε να μιλήσετε. Να είστε σύντομος. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, να πω ότι στην ε, ομιλία μου λόγω χρόνου εστίασα στο δεύτερο τμήμα. Στο πρώτο τμήμα εκεί γίνεται λόγος για το πλαίσιο και για την χρηματοδότηση. Αν λοιπόν δούμε πιο συγκεκριμένα τις παραγράφους 17 και 25, εκεί γίνεται περιγραφή των υποδομών, των αναγκών και της διαθεσιμότητας των κονδυλίων. Και στον πίνακα υπαριθμών 2 βλέπουμε ε, εκταμείευση κονδυλίων για την περίοδο ε, μέχρι το 2020 από το ε, τα Συνοχή, από το Μάρκο Πόλο, από το FP7, από το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ε, τα οποία εξηγούν ε, το τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά τα κονδύλια. Κυρίως όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει σελίδα 39 παράγραφος 72, εκεί ε, λέμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε προτεραιότητες, σε τομείς με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ε, κάθε κονδύλι περιγράφεται συγκεκριμένα σε εκθέσεις. Σας είπα ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια ειδική έκθεση για τις μεταφορές. Η χρήση των κονδυλίων σε αυτή την έκθεση αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια. Εδώ είναι απλά η περίληψη όλων αυτών. Αυτά που σας έφερα είναι η περίληψη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχουμε άλλη μια ειδική έκθεση. Ο κύριος Τσέλερ παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ ε, θα ήθελα να πω το εξή. Η συγγήτρια, η συνάδελφός μου, η Κλάουντια Σμιτ, είναι η συγγήτρια, η συνάδελφός μου. Όχι, πρώτα να κλείσουμε το 9 και μετά το 10. Για το 9. Να σας πω ότι όπως είπε και η Κομισιόν έχουμε ένα πολύ καλό στρατηγικό σχεδιασμό για την διασύνδεση των μεταφορών. Οι ε, νομικές προϋποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και ελπίζω ότι <clears throat> αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιτέλους, ε, όπως είπε και η κυρία Γιάλα Σέντερ, να προσκρούσουν σε γόνιμο έδαφος στα κράτη-μέλη και να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια επέκταση του δικτύου των μεταφορών, κυρίως ε, να βελτιωθούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Ελπίζουμε, εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει το Brexit. Αν όμως τελικά αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία, θα δούμε τι ακριβώς ε, θα σημαίνει το να ε, καταρρεύσουν δομές ε, που μέχρι τώρα χρηματοδοτούν το μια χαρά. Και θα δούμε τότε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την οικονομία και για την κινητικότητα των ανθρώπων. Και ίσως τότε κάποιοι να σκεφτούν ότι θα πρέπει να ισχύει ακριβώς το αντίθετο αυτά τα οποία μας είπε και το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή οι ε, δυνατότητες ε, που υπάρχουν έτσι ώστε να ε, επιτύχουμε ένα δίκτυο, όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν να τύχουν της σωστής εκμετάλλευσης. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης που αφορά στα δικαιώματα των επιβατών. Το λόγο έχει ο κύριος Πουφάν. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες μου και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ε, επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ σε όλους ε, καλή χρονιά 2019. Είναι μεγάλη τιμή που έχω να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση παριθμό 30 2019 με τίτλο «Οι επιβάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαιώματα αλλά δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους». Πού βασιστήκαμε στην εφαρμογή του πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών και αρθρώνεται γύρω από διάφορους κανονισμούς που διέπουν ε, τις εναέριες μεταφορές, τις σιδηροδρομικές, τις ε, οδικές με λεωφορεία και τις ε, πλωτές. Υπάρχουν δικαιώματα για τους επιβάτες, αλλά παραμένουν μεγάλα προβλήματα στην υλοποίησή τους όταν τα διεκδικούν τα δικαιώματά τους αυτά θα ήθελα να σας μιλήσω για τρία σημαντικά προβλήματα, τα σημαντικότερα, και να σας αναφέρω και τις βασικές συστάσεις της έκθεσής μας. Καταρχάς, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής γεγονός. Ε, οι εργασίες μας βασίστηκαν στα θεμελιώδη λεγόμενα δικαιώματα των επιβατών, δικαίωμα στην πληροφορία και δικαίωμα στην ε, συνέχεια που δίνεται στο πρόβλημά τους και στην αποζημίωση. Είναι πολύ διαφορετική κατάσταση ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Ε, τα δικαιώματα των ε, επιβατών δεν είναι πάντα σαφή για τους ίδιους τους επιβάτες, αλλά ούτε και για τις μεταφορικές εταιρείες, ε, ούτε για τις εθνικές αρχές που έχουν επομιστεί με το σεβασμό ε, αυτών των δικαιωμάτων. Ας πούμε, το δικαίωμα να ασχοληθεί κάποιος μαζί σου όταν διακόπτεται το ταξίδι σου ε, δεν είναι σαφώς ορισμένο στον κανονισμό. Πολλές φορές οι εταιρείε ε, αποφασίζουν μόνες τους ε, τι προστασία θα μας δώσουν εμάς ως επιβάτες όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μεταφορά. Οι επιβάτες όμως, αν γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους, θα εξισορροπήσουν ξανά την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια ε, του ελέγχου δυστυχώς ε, φάνηκε ότι η ευαισθητοποίηση των επιβατών είναι της τάξεως του 40% αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχο επίπεδο με ε, αυτό που είχε διαπιστωθεί πριν από μία τετραετία. Επειδή είναι το πλαίσιο περίπλοκο, δημιουργήθηκε ένα νέο είδος οργανισμού παραπώνων για εξοδικαστική και επίλυση διαφορών. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει αδιαφάνεια στο πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Σήμερα ένας επιβάτης δεν έχει καθόλου ενημέρωση για το λόγο της καθυστέρησης της πτήσης ας πούμε ή του ταξιδιού του ούτε ε, τι δικαιώματα έχει και τι, ε, από τι υποφελούνται άλλοι επιβάτες ε, που έχει διακοπή για τους ίδιους λόγους στο ταξίδι τους. Το ίδιο ισχύει δυστυχώς και με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές για την αποζημίωση για φέρει τον επαναπατρισμό ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια είναι δυνατόν, για να μην πω ότι είναι συχνό, να παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών, των επιβατών και βρήθη ε, των ανισότητα στη μεταχείριση έκθεσή μας. Πέντε είναι οι συστάσεις που απευθύνουμε γενικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνήσανε ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πρώτον, ε, προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τα 10 θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών προστατεύονται στα τέσσερα μέσα μεταφοράς και να δούμε ή δυνατόν ε, πώς μπορούν να μειωθούν οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφοράς. Στη συνέχεια ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει νέες κατευθυντήριες γραμμές με κατώτατα πρότυπα για ε, την ενημέρωση των επιβατών σε περίπτωση που ε, έχει προβλήματα η ε, μετακίνησή τους και τι δικαιώματα έχουν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους ή ακόμα και η προσφυγή σε, άλλα, σε άλλο μεταφορέα. Η τρίτη σύσταση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, λανσάρει σε στενό συντονισμό μαζί ε, με τα κράτη-μέλη ε, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το 40%. Τέταρτη σύσταση έχει να κάνει με την αδιαφάνεια. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει κατώτατα πρότυπα παροχής βοήθειας. Αυτή τη στιγμή Το μόνο που δίνουν ως βοήθεια στους επιβάτες είναι ε, ότι θα τους επιστρέψουν κάποια χρήματα κάποια στιγμή. 40 ευρώ ε, προτείνουμε εμείς ε, για τους επιβάτες. Και για, επίσης το επόμενο 48 ώρο ε, όταν υπάρχουν επιπτώσεις λόγω καθυστερήσεων ή ακυρώσεων, θα πρέπει οι αρμόδιοι ε, οργανισμοί, οι εθνικοί οργανισμοί να αναλύσουν ε, τις πρακτικές των μεταφορέων. Αν αναγνωρίσει ο μεταφορέας ότι η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε δικό του σφάλμα, τότε περιμένουμε αυτόματα να αποζημιώνει με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Και τέλος καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις έτσι ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των εθνικών οργανισμών που είναι αρμόδιες για τα δικαιώματα αυτά και να έχουν και εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει όλη αυτή την προσπάθεια. Θα σταματήσω εδώ την παρουσίασή μου. Είμαστε στη διάθεσή σας, οι συνεργάτες μου και εγώ, για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πουφάν. Ο κύριος Τσέλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εδώ πάλι είναι η γνωμοδότηση της συναδέλφου μου Κλάουντια Σμιτ, αυτή που σας παρουσιάζω. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την ε, ε, εκτεκτή έκθεση αυτή ειδική έκθεση και τον κύριο Πούφαν και τους συνεργάτες του. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί ε, ραγδαία η κυκλοφορία των επιφανών και πραγματικά ήταν ορόσημο ύπαρξη των δικαιωμάτων των επιβατών γιατί αν ε, δούμε περί τίνος πρόκειται και ποια είναι τα συμφέροντα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποζημιώσεις. Βέβαια ε, πολλά από όσα λέει ο κανονισμός και η νομοθεσία ε, χωράνε ευρύ ερμηνεία. Τι θα πει ενημέρωση, υποστήριξη, βοήθεια, ε, πλαισίωση και γιατί θα γίνει, και, σημαίνει ότι με άλλο τρόπο θα μεταφερθεί ο επιβάτης από εκείνο που είχε προβλέψει αυτό, Εμποδίζουν τους επιβάτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στην αρμοδιότητα των εθνικών οργανισμών ε, υλοποίησης και προβλέπονται και πολλές εξαιρέσεις στην νομοθεσία. Αυτά όλα περιορίζουν τα δικαιώματα των επιβατών. Η κυρία Σμίτ είναι συχνά επικριτική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα θέλει να την επενέσει. Η εποπτεία και παρακολούθηση ε, των, ε, της υλοποίησης και εφαρμογή των δικαιωμάτων των ε, επιβατών βοήθησε να γίνουν οι κανονισμοί πιο διαφανής και πιο εύληπτοι. Βέβαια δεν έχει εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εναρμόνιση της υλοποίηση και της ερμηνείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ακριβώς επειδή στερείται αυτή τη στιγμή εντολή για να επιβάλλει τα δικαιώματα έχει συμφωνήσει με τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου η κυρία Σμίτα αναφέρεται στην αλλαγή, τροποποίηση του κανονισμού και ρωτάει μετά την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού, πώς βλέπει τις ε, πιθανότητες ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιωθούν ε, τα δικαιώματα αυτά και να επιβάλλονται καλύτερα. Τι γίνεται με τις ενημερωτικές θηρίδες και ποια δυνατότητα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν ε, διευρυνθεί η εντολή της να ε, βελτιώσει την προστασία και τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Και ευχαριστή κυρία Σμιτ για την απάντηση. κύριος Ρόιτας. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους ε, για αυτή την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της αυτήν την έκθεση και δέχεται τις συστάσεις. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος χώρος ε, σε όλο τον κόσμο που προσφέρει πλήρη δικαιώματα στους επιβάτες και προχωρήσαμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε εξυγχρονίσει τους κανονισμούς το 2013. Έχουμε ε, και μία άλλη πρόταση που κατατέθηκε το 2017 για τα δικαιώματα των επιβατών. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν γρήγορα με αυτές τις δύο προτάσεις που έχουν ως στόχο να επιτευχθούν οι προτάσεις, οι συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Απαντώντας σε αυτά που λέει η κυρία Σμίτ, θέλω και εγώ να πω ότι βεβαίως ε, εμείς θεωρούμε ότι ο έλεγχος είναι μια ευκαιρία ε, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή προστασία ε, των επιβατών και να δρομολογηθεί ε, απλούστευση των περίπλοκων μηχανισμών και τελικά να συμφιλειώσουμε οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο τον κλάδο με τους επιβάτες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με δύο προτάσεις ε, οι οποίες ε, τώρα βρίσκονται στη διαδικασία της ε, συναπόφασης. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ανασταλεί ο κανονισμός του 2013 λόγω της διαφοράς απόψεων για το Γιβραλτάρ. Μπορεί όμως να επανέλθει αυτός ο κανονισμός Βεβαίως εμείς ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτή τη νέα πρόταση που σας είπα για τα δικαιώματα των επιβατών. Θέλουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον θα ήθελα βέβαια να απευθυνθώ και στον κύριο Τσέλα και στην κυρία Σμιτ και να τους πω ότι το 19 θα ε, καταθέσουμε μία μελέτη ως συνέχεια αυτή της έκθεσης. Ε, θα την επεξεργαστούμε αυτή τη μελέτη για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να παγιώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών με έναν τρόπο που να μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Ε, θέλουμε, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα. Αυτό που θα εξετάσουμε επίσης είναι να έχουμε και το δικαίωμα δικαίωμα της ε, πρωτοβουλίας για να καταθέσουμε προτάσεις ε, στις ε, προκλήσεις που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο. Είμαστε πολύ θετικοί και θέλω να σας πω ότι και εμείς από δικής μας πλευράς θέλουμε να επενέσουμε το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ καλή έκθεση που κατέθεσε επί του θέματος. ο συνάδελφος φάει για να ολοκληρώσει και μετά ε, ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι στο μέλλον ενδεχομένως η εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσαρμοστεί ανάλογα. Πιστεύω πάντως ότι ε, ο έλεγχος αυτός μας επιτρέπει όντως να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να τελειοποιήσουμε τα νέα νομοθετικά μέτρα και να καταφέρουμε να καλύψουμε με ένα νέο κανονισμό και τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών. Στεργαστήκαμε πάντως πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξέρετε, κι εγώ τυχαίνει να είμαι επιβάτης μερικές φορές και ειλικρινά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά Πώ έχουν τα πράγματα, τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν όταν πρέπει για παράδειγμα να αλλάξει κανείς αεροδρόμιο. Δεν είναι πάντα εύκολο στην περίπτωση αυτή να βρει κανεί ε, μία άλλη πτήση. Προκύπτουν επίσης ιδίως στην περίοδο των Χριστουγέννων πολλά προβλήματα. Μία φορά χρειάστηκε και εγώ να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο πρόβλημα. Είχα μία πτήση σε δύο σκέλη και στο δεύτερο σκέλος έπρεπε να διασχίσω τον Ατλαντικό. Ξέρετε ότι σε τέτοιες πτήσεις, αν χάσει κανείς την πρώτη του πτήση, το πρώτο σκέλος, είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρει να μεταβεί όντως γρήγορα στις ΗΠΑ, στο συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα το οποίο έθεσα. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές φορές είναι πιο εύκολο να πάει κανείς με το αυτοκίνητο στην Φραγκφούρτη και από εκεί πέρα να πάρει μια απευθείας πτήση. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει κανείς στο τελικό του προορισμό. Τουλάχιστον εγώ αυτό σκέφτηκα για την περίπτωση αυτή που χρειάζεται να αντιμετωπίσω. Αφορά αυτό όλους μας ε, και αν κάνουμε εδώ μια μικρή έρευνα, ε, και εγώ ας πούμε ε, πήγαινα στην Τσοχοσλακία, τελικά κατέληξα στη Βαρσοβία, μπρος πίσω, δεν ήταν δυνατόν να προληπτήσει πολύ κνευριστικό αυτό να βρίσκεται κανείς μπλοκαρισμένο κάπου χωρίς να έχει καμία απολύτω πληροφόρηση. Ο κύριος ε, Τσέλερ. Ε, ε, εδώ προσυπογράφω, επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ, έχω και αντίστοιχη εμπειρία αποκομίσει. Όπως ήδη είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέτος είναι ιδιαίτερη χρονιά, προεκλογική, που μας ρωτάνε σε τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενίσχυση των επιβατών αεροπλάνων και ε, λεωφορείων ε, και σιδηροδρόμων είναι κάτι το οποίο δεν ε, τονίζεται συχνά. Βεβαίω το καλύτερο είναι εχθρό του χαλού. Πάντα υπάρχει καλύτερο. Έκανε κάποια συστάσει στο ελεγκτικό συνέδριο. τις δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πραγματικά η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών και η άσκησή τους είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Ελπίζουμε να προχωρήσει και ε, να μπορέσουμε έτσι αναλόγως να το τονίσουμε και φέτος στην προεκλογική εκστρατεία. Ωραία. Τελείωσε και αυτό το θέμα της μέρης σας διάταξης. Ευχαριστώ. 11. Διάφορα. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Θέλω να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 21 του μηνός, στις 3 εδώ στις Βρυξέλλες. Καλά να περάσετε μέχρι τότε. σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Λήξη συνεδρίασης.